Right. Good morning everyone. Good morning ladies and gentlemen. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. I would like to welcome you all to our θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ε, πρώτη μας ε, συνεδρίαση μετά τις καλοκαιρινές ε, διακοπές. Ελπίζω να περάσατε καλά, να χαρήκατε τον καλοκαιρινό ήλιο. Και τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το σχέδιο ημερησίας διάταξης. Έχουμε την έγκριση της ημερησίας διάταξης υπό το σημείο 1. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνεται. Δεν έχω ανακοινώσει εγώ ως πρόεδρος προς το παρόν. Επομένως, μπορούμε ήδη να περάσουμε στο σημείο 3. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό της 2019, όλα τα τμήματα. Ο κύριος Μπενιφέη, ο συνάδελφος, είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης. Καλώς ήλθατε και θα μπορούσαμε να περάσουμε απευθείας στις ψηφοφορίες εκτός αν ο εισηγητή θέλει το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Επομένως, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με τον κατάλογο ψηφοφοριών για την δημοσιονομική διαδικασία. Και πώς να το ανακοινώσω. Για να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 536. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5237 υπέρ. Κατά. Αποχές. 5158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51-59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52-01 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65-29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52, 33 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 52, 32 αποσύρεται. Πάμε στην 52, 31 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβεστική 1 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 52, ε, 03 εγκρίνεται. 51, 63 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 51, 64 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 52-35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51-66 υπέρ, κατά, αποχές. Λοιπόν, για να ελέγξουμε για πρώτη φορά την 51-66, έρχεται η ψηφορία. The Λήξη απορρίπτεται με 18 αποχές, 24-8. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 52-05 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 51-72 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 5172. Λήξη. 47 προς 4, ξεκάθαρο αποτέλεσμα, 52.06 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51.73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51.79 εγκρίνεται, 51-50 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται, 51-90 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται, συμβαστική 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 52-08 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 51-71 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 5228 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 52-30 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-13 υπέρ κατά αποχε εγκρινεται εγκρίνεται. 52-14 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Καταπίπτει. Επόμενη 51-51 υπέρ κατά εποχές. Να ελέγξουμε την 51-51 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 28 προς 22. 52-15 υπέρ κατά εποχές. Εγκρίνεται. 52-16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, καταπίπτει αυτή. Είναι συμβεστική 8, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 9, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-19, υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. εγκρινεται Εγκρίνεται ξεκάθαρα. 52-20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52-21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 κατά πίπτη. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε μια ψηφοφορία σε blog 5. Τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Στη συνέχεια πάλι έχουμε ψηφοφορία ομαδική από την 5175. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελος 5176 υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται. Αυτά. We then come to... Να περάσουμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2019, όλα τα τμήματα, ο Μπράντο Μπενιφέ και πάλι είναι εισηγητής. Θέλετε να πείτε κάτι τώρα, όχι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 4, άρχεται τη ψηφορία. Λήξη. Ξεκάθαρο αποτέλεσμα. 5. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν ανακοινώσα το αποτέλεσμα. 26 προς 7 ή κάτι τέτοιο. Και 21 αποχές. Πάμε στην τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 ως 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 44 καταπίπτει, 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη γραμματότηση όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Και οι 56 ψήφισαν. Τέλος. 43 υπέρ, 5 κατά, 8 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και σας ευχαριστούμε για την καλή δουλειά. So. Λοιπόν, είναι εδώ ο Υπουργό Εξωτερικών. Θα σας ζητήσω να παραμείνετε όλοι στην αίθουσα. Σε λίγα λεπτά θα ε, έρθει και ο Υπουργός.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 So, ladies and gentlemen, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες ε, της Επιτροπής μας. Έχουμε τη συζήτηση ε, για την έκθεση πρόοδου των ε, τρίτων χωρών. Έχουμε λοιπόν μαζί μα τον Νικόλα Δημητρόφ, Υπουργό Εξωτερικών τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονία, τον οποίο καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μα. Να χαιρετήσουμε θερμά και την νέα πρέσβυρα ε, τη Μακεδονία, κυρία Γκρουπόφσκα. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα και καλή επιτυχία σα ευχόμαστε. Ο κύριο Δημητροφ είναι Γνωστό, βέβαια εδώ και στον ε, πολιτικό βίο της χώρας του. Έχουμε υψηλέ προσδοκίε από τη νέα κυβέρνηση μετά το 2017, μετά από μια μακρά και άρευ προηγουμένου πολιτική κρίση. Πλέον, σε αντίθεση με το παρελθόν, ε, ξαναφέρατε τη χώρα σας ε, ανάμεσα σε αξιόπιστους εταίρους. Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις μετά την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ. Ε, πολύ εντυπωσιακή εξέλιξη μετά την τελευταία σας παρουσία τον Οκτώβριο του 2017. Οι ε, προσπάθειε σας έχουν αναγνωριστεί και από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΟΗΕ ξεκινούν οι προσπάθειες για την ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ το, και οι διαπραγματεύσει θα ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι. Να σας δώσουμε λοιπόν το λόγο για να μας δώσετε την εικόνα στη χώρα σας από τη δική σας σκοπιά ε, πώς βλέπετε τις εξελίξεις εν ώψη και του επερχόμενου δημοψηφίσματος. Εμείς εδώ, με μεγάλο ενδιαφέρον, ε, θα ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μακάλιστερ. Πάντα είναι μεγάλο προνόμιο για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Αυτή τη φορά ήταν ε, εύκολο το ταξίδι, ομαλή μετάβαση. Ελπίζω ομαλή να είναι και η μετάβαση και το ταξίδι που περιμένει τη χώρα μου από τώρα μέχρι και τον επόμενο Ιούνιο, ελπίζω. Και να λήξει το 2019 με μια διακυβερνητική συνδιάσκεψη. Θα είμαι σύντομος, θα επικεντρωθώ στα κέρια ζητήματα για να έχουμε και περισσότερο χρόνο για ανταλλαγή απόψεων περιμένω να ακούσω και τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εξάρω τη σοφία του οίκου της Δημοκρατίας εδώ, της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι ε, συνεχής ε, η προσήλωσή σας σε ό,τι αφορά τη στήριξη του μέλλοντος των Βαλκανίων. Και μάλιστα αυτό σε όλο το πολιτικό φάσμα και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν όλοι και οι υποψήφοι, οι υποψήφιες χώρες, ε, αν είχαν ακολουθήσει αυτές τις συμβουλές σας ε, ε, σε όλο το φάσμα των ετών. Είχαμε και τον διάλογο του Ζαν Μονέ και το Σεπτέμβριο θα έχουμε τη συνέχιση της διαδικασίας, προβλέπουμε σε αυτό. Από κοινού διοργανώνουμε και μία συνδιάσκεψη ε, το Σεπτέμβριο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάλι στα Σκόπια. Φέρνω καλές ειδήσει, το οποίο μπορεί να προκαλεί έκπληξη, γιατί είναι δύσκολη η καιρή ε, που περνούμε και στην Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής. Αλλά το καλύτερο είναι να δούμε από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Ξεκινήσαμε την 1η Ιουνίου του 2017. Λίγες μόνο ημέρες μετά από την πιο μελανή σελίδα ε, στην ιστορία μας όταν ένας ε, άνθρωπος ε, επιτέθηκε στο κοινοβούλιο μας. Υπάρχουν ζητήματα υπήρχαν στο παρελθόν ζητήματα στη χώρα μου, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, την ελευθεροτυπία. Κάποιοι αποφάσισαν μάλιστα να μην ε, ε, μεταφέρουν ε, στα, στην τηλεόραση και στον τύπο την υπόθεση αυτή με την επίθεση στο Κοινοβούλιο ή με τις υποκλοπές ή με τη διαφθορά, γιατί είχαμε και τέτοια περιστατικά. Τώρα έχουμε κάνει μία στροφή 180 μοιρών και Προσπαθούμε να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία, αυτή την οπισθοδρόμηση, να ανοικοδομήσουμε τη δημοκρατία μας, ίσως ακόμα παραπέρα, γιατί έχουμε μια όρημη κοινωνία πλέον. Ε, υπάρχει θυμός στην κοινή γνώμη και πλέον ε, υπάρχει μεγαλύτερη τόλμη σε ό,τι την κοινωνία των πολιτών. Επομένω, μάθαμε ότι έχει νόημα το να λαμβάνει κανείς θέση και να την δημοσιοποιεί. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν υπήρξε μια διαρροή των οικονομικών αποζημιώσεων που λαμβάνουν τα μέλη της ε, ε, εκλογικής επιτροπής, το, η κοινή γνώμη ε, αντέδρασε με τόσο νητικό τρόπο που αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα της κρίσης, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι οι πολίτες μας έχουν αντιλήσει ένα σημαντικό δίδαγμα. Επιπλέον τη στρατηγική μας για το κράτος δικαίου και με τους νέους νόμους που έχουμε ψηφίσει στο Κοινοβούλιο, πλέον αυτό που έχει σημασία είναι η εφαρμογή τους. Έχουμε διαδικασίες που, ε, και υποθέσεις που συνδέονται ε, με τον κατήγορο και συνεχίζεται η διαδικασία κατά των ε, των όσων σχεδίασαν και υλοποίησαν την επίθεση στο Κοινοβούλιο πέρσι. Ξέρω ότι εδώ προέρχεστε από διαφορετικέ οικογενειακές, πολιτικές οικογένειες. Μπορώ να σα πω ότι η πολιτική κρίση ε, στην Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν ένας εφημισμός για μια ε, κρίση ατιμορρησία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια των συνηθισμένων πολιτικών ανταγωνισμών μεταξύ αριστεράς και δεξιάς για μας ε, ο αγώνας ήταν να σώσουμε τη δημοκρατία μεταξύ του ορθού και του λάθους λοιπόν, του δίκαιου και του άδικου. Η πολιτική κινητοποίηση λοιπόν δεν ήταν μόνο μεταξύ εθνοτικών ή μάλλον που να ενώνει εθνοτικές ε, ε, μειονότητες αλλά και πολιτικές απόψεις. Στα μέσα μαζική ενημέρωση η κατάσταση βέβαια είναι τελείω διαφορετική, σαν να μιλάμε για διαφορετική χώρα. Ε, υπάρχουν συζητήσει που είναι υγιεί σε μια δημοκρατική κοινωνία. Πριν από τι εκλογέ του 2016, για μια σειρά ετών δεν υπήρχε συζήτηση, πολιτικός διάλογος μεταξύ πολιτικών αντιπάλων πριν από τις εκλογές. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική μα πολιτική και τι διεθνεί μα σχέσει, έχουμε πέντε γειτονικέ χώρε. Είχαμε ζητήματα με πολλέ από αυτέ. Δύο ήταν τα μείζωνα ζητήματα με τα δύο, ε, τις δύο γειτονικές μας χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνε φίλοι μας και οι φίλοι μας από την Βουλγαρία. Από την αρχή της ε, κυβέρνησή μας. Εμείς ε, ήρθαμε σε επαφή με τους συναδέλφους μας. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή με μεγάλη ιστορία, αλλά δεν ασχολείται αρκετά με το παρόν και το μέλλον της. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, ούτε την ιστορία μας. Μπορούμε όμως, εάν επικεντρωθούμε σε αυτό, να διαμορφώσουμε το κοινό μας μέλλον, που είναι και ευρωπαϊκό. Υπήρξε λοιπόν μία συμφιλίωση και μία ενοποίηση μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό κάναμε. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σούμαν είχε πει ότι η Ευρώπη δεν θα οικοδομηθεί ε, με τη μία ή με βάση ένα ενιαίο σχέδιο, αλλά θα οικοδομηθεί μέσω συγκεκριμένων επιτευμάτων που θα δημιουργήσει, δημιουργήσουν μία de facto αλληλεγγύη. Αυτό που έκαναν η Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Βουλγαρία και η Ελλάδα ήταν ακριβώς αυτό. Συγκεκριμένα επιτεύγματα που δημιουργούν μία de facto αλληλεγγύη. Και θα ήθελα εδώ, ενώπιόν σας και δημοσίως, να εκφράσω τα θετικά μου σχόλια ε, για τις ηγεσίε Σόφιας και Αθηνών, που κατέστη σαφής κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, κάτι που στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θα κάνω πολλές ακόμα παραθέσεις, αλλά αυτή είναι μια σημαντική, γιατί θα ήθελα να τονίσω το μέγεθος και τη σημασία αυτής της επιτυχίας. Γιατί δεν ήταν πρόκειται μόνο για μια επίλυση μιας ε, τυπικής ε, διμερούς ε, διαμάχης στα Βαλκάνια. Ένας Γάλλος γενοούμενος κάτοχος του βραβείου Νόμπελ που ηγείτο της Επιτροπής Κάρνεγκη που είχε πάει στα Βαλκάνια για να διερευνήσει την κατάσταση το 1914. Και παραθέτω λοιπόν οι πραγματικοί υπέτη είναι αυτοί που εθυσιάζουν το γενικό συμφέρον για το προσωπικό του συμφέρον. και επακολουθούν μια στήρα πολιτική ε, διαμάχης. Στην πράξη δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει διέξοδος ούτε για τα μικρά κράτη, ούτε για τις μεγάλες χώρες, παρά μόνο ε, μέσω της ένωσης και της συμφιλίωσης. Αυτό συνέβη λοιπόν πραγματικά τους τελευταίους 14 μήνες στην περιοχή μας. Χαίρομαι που πολλά κράτη-μέλη, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, αναγνωρίζουν πλήρως αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, δεν θέλουμε χάρες, δεν θέλουμε μια πολιτικοποιημένη διαδικασία ένταξης, δεν θέλουμε να ανταμυφθούμε μόνο για το πολιτικό θάρρος που έχουμε επιδείξει και για το όραμα που έχουμε για το μέλλον και για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Όλες οι χώρες θα πρέπει να κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους, βάσει των κριτηρίων της Κοπεχάγης. Και η υλοποίηση του σχεδίου 369 μας φέρνει σε θέση και δείχνει μάλλον ότι έχουμε σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο στους εννέα τομείς ε, που εξετάζει κατά κύριο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε σημειώσει πρόοδο ε, σε πέντε από τους εννέα αυτούς τομείς. Και προχωράμε. Εν συντομία θα ήθελα να αναφερθώ και στην ευρύτερη περιφέρεια. Γιατί σίγουρα θα τα συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Μίλησα για το κράτος ε, δικαίου, ε, για την δημοσιοδιοίκηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, και τη μεταρρύθμιση του κλάδου των μυστικών υπηρεσιών. Ξέρουμε ότι οι συζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή επικεντρώνονται και σε άλλα ζητήματα. Πρόσφατα έγινε λόγος ε, για τον διάλογο μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου. Εάν θέλουμε ειρήνη στα Βαλκάνια, δείτε το, τη δεκαετία του 90, κέρδισε το ευρωπαϊκό όραμα. Όλοι προχωρήσαμε, όλοι εργαστήκαμε σκληρά για να βρούμε την ισορροπία και συμμεριζόμαστε ένα όραμα όπου η περιφέρεια εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου τα σύνορα δεν έχουν πια τόση σημασία. Το γεγονός ότι ε, τίθεται αμφιβόλο σε έναν βαθμό αυτό το όραμα και έχουμε την επιστροφή γεωπολιτικών ανταγωνισμών στα Βαλκάνια, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ε, έλλειψη ε, προόδου και δυναμικής, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την ανταξιακή διαδικασία. Δεν μπορώ εγώ να δω άλλο όραμα για μια βιώσιμη ειρήνη, δημοκρατία και ευημερία στην περιφερειά μας. Πρέπει να επικεντρωθούμε και να δώσουμε την απαραίτητη ενέργεια, να επενδύσουμε στην ενταξιακή διαδικασία. Όποτε υπάρχουν επιτυχίες, θα πρέπει να ανταμείβουμε τις ε, υποψήφιες χώρες. Όποτε υπάρχει οπισθοδρόμηση θα πρέπει να τις ε, κατονομάζουμε. Και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να εντάξουμε πραγματικά αυτή την ε, περιοχή. Γιατί συχνά σκεφτόμαστε ότι τα Βαλκάνια βρίσκονται στην περιφέρεια. Είναι μια νησίδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες φορές βρίσκεται έχει ίσονα σημασία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, αλλά βρίσκεται στο κέντρο. Και από τη δικασία του 2015 και του 2016 αυτό διαφαίνεται. Και εκείνα τα γεγονότα δείχνουν γιατί αυτή η περιφέρεια είναι τόσο κρίσιμη σημασία για την ε, ειρήνη και ευημερία. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ε, αγορά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Τρία τέταρτα των ε, ε, ξένων επενδύσεων προέρχονται από την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αλληλεπίδραση και από οικονομικής άποψης, πολιτικής και από πλευράς ασφάλειας. Το τελευταίο για τη σημερινή κατάσταση, για το δημοψήφισμα, είναι ιστορικής σημασίας η σημερινή συγκυρία όταν ανεξατοποιήθηκε η Δημοκρατία της Μακεδονίας ήμουν 18, του χρόνου γίνομαι 46 και είναι η δεύτερη ευκαιρία για τη γενιά μου να διασφαλίσει ότι η χώρα μας ε, θα περάσει αυτή την γραμμή της σιγουριάς. Εδώ και πολύ καιρό περιμένουμε έξω από την είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Για να έχουμε μια επιτυχή χώρα στα Βαλκάνια, πρέπει όλη η περιοχή των Βαλκανίων να πετύχει. Όλοι είμαστε φυσικοί σύμμαχοι. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι μια, ένας ανταγωνισμός μεταρρυθμίσεων Ποιο έχει τη μεγαλύτερη ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης, Ποιο έχει ε, πιο καλή δικαιοσύνη, περίθαλψη, παιδεία. Ο ανταγωνισμός τώρα για την ιστορία. Ποιος ε, είναι ο λαός με τη μεγαλύτερη ιστορία ή το έθνος με τη μεγαλύτερη ιστορία. Ποιος έχει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ε, στην ιστορία του δεν είναι υγιής και παραγωγικός ανταγωνισμός. Και παρότι όλοι είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι αυτή η γενιά μπορεί να είναι περήφανη για τα επιτεύγματά της σήμερα και αύριο. Και αν δεν τα καταφέρουμε, όλα τα ταλέντα μας ε, θα φύγουν από τη χώρα μας και θα πάνε στις δικές σας. Για να μην λοιπόν η νέα γενιά στην πατρίδα μας, θα πρέπει η Ευρώπη να έρθει, να φέρουμε την Ευρώπη στην περιφέρεια και στη χώρα μας. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε αυτό. Θα κερδίσουμε το δημοψήφισμα. Κατά παράδοση κάνουμε σοφές επιλογές όταν μας τίθενται δύσκολα ερωτήματα. Και θα μπορούσε βέβαια η πολιτική κατάσταση να είναι καλύτερα από πλευράς ευθύνης, γιατί ορισμένοι από τους πολιτικούς μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τις πράξεις του παρελθόντος και κάποιοι δεν αντιμετωπίζουν την ευθύνη του μέλλοντός μας. Αυτά είναι δύσκολα ερωτήματα. Για κάποιους αυτό θα είναι πολιτική αυτοθυσία, αλλά το δημοψήφισμα δεν έχει να κάνει με τα πολιτικά κόμματα, δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς, δεν είναι θέμα ε, αν θέλει κανείς αυτή την κυβέρνηση ή όχι. Πρόκειται για το μέλλον της χώρας. Πρόκειται για την οικοδόμηση ε, φιλίας, σχέσεων φιλίας σε μια περιοχή που τις χρειάζεται. Μένω εδώ και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Δημητρόφ για την παρουσίαση για τις πολιτικές απόψεις κατά τον χρόνο 16 λεπτών Τώρα, πότε έρχεται στην, στην Επιτροπή μας, πολλοί συνάδελφοι έρχονται και πολλοί ενδιαφέρουν να πάρουν το λόγο. Έχουμε έναν αριθμό ρεκόρ ετοιμάτων και έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Έχουμε ήδη 17 συναδέλφους. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι όσο πιο δίκαιος γίνεται σε, όλα, σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Αυτό που προτείνετε να του ακούσουμε όλου ή να το μοιράσουμε στα δύο. Να το μοιράσουμε στα δύο. Και όταν θεωρείς ότι είναι αρκετά τα ερωτήματα, τότε μπορούμε να διαγράψουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το ΕΛΚ. Ο κύριος Πρέντα. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την ομιλία σας. Θα ήθελα να πω εντάχει δύο πράγματα. Πριν ε, τέσσερα χρόνια είμαστε κάπως ε, διστακτικοί στα Δυτικά Βαλκάνια, απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια και η πλειοψηφία έλεγε ότι δεν θα γίνει η διεύρυνση από αυτή τη θητεία όμως έχουμε δει αλλαγές ε, τους τελευταίους μήνες, ε, καταρχήν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε και στο επίπεδο Συμβουλίου θα κερδιθεί εμπιστοσύνη σε σχέση με τα γεγονότα στα Δυτικά Βαλκανία, γιατί η συμφωνία μεταξύ Μακεδονίας και Ελλάδας δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορούν να μετακινηθούν προς την ορθή κατεύθυνση τα Βαλκάνια. Είναι πολύ καλή είδηση αυτή και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα δύο μέρη και τους Μακεδόνες και τους Έλληνες ε, στην επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Christian. Ευχαριστώ. Περνάμε στο λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την πρέσβη της Γεωργικής Δημοκρατίας της ε, Μακεδονίας. Είναι μεγάλη ε, χαρά για μας. Συμφωνία που επιτεύχθη γιατί αυτό καθιστά όλη τη διαδικασία ε, πιο λογική. Θεωρώ ότι θα είμαστε εξίσου χαρούμενοι μετά την 30 Σεπτεμβρίου και μετά το δημοψήφισμα. Ποια είναι η αξιολόγησή σας σχετικά ε, με το δημοψήφισμα. Δεύτερο ερώτημα. Ξέρω ότι πολλοί έχουν ε, επενδύσει πολύ στα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος την, ε, και ότι θα την επανφέρει σε μια κατάσταση ανασφάλειας, όπως και πριν. Έχει να κάνει αυτή η αντίληψη με κάποιες εξτρατείες που ε, γίνονται εκτός ε, της χώρας και πιστεύετε ότι ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσουν ε, το αποτέλεσμα του ψηφίσματος. Θεωρείτε ότι οι παράγοντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν ρόλο σε αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό στη Μακεδονία. Ευχαριστώ τον Νίνο. Τσάρλσταν και το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλώς ήρθατε κύριε Δημήτροφ. Είμαι ιδρυτή των φίλων τη ε, Μακεδονία και υποστηρίζω τη χώρα εδώ και 20 χρόνια από αυτή την επιτροπή. Παράλληλα όμω είμαι και φιλέλληνα σε όλα τα θέματα, εκτό από το θέμα τη ονομασία τη χώρα σα και δείχνω συμπάθεια προ τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα σα την εθνικό, εθνικό διαχωρισμό, του πολέμου κτλ. Τώρα όμω ε, διαφαίνεται ένα πιο λαμπρό μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνησή σα πρέπει να δεχτεί τα συγχαρητήρια για την ιστορική σημασία σε απόφαση για την ονομασία και φυσικά έχετε την πλήρη στήριξη της ε, πολιτικής μου παράταξης και ευχόμαστε να εξπεράσετε το τελευταίο εμπόδιο της 20 Σεπτεμβρίου και του δημοψηφίσματος θα σας οδηγήσει ε, στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης ε, προσχώρηση και στο ΝΑΤΟ. Ελπίζω ότι θα εισέλθετε σε μια περίοδο σταθερότητας μετά από τη συμφωνία με το Κόσοβο, το Κοσοπέδιο και την Σερβία. Και το καλό είναι επίσης ότι οι μετασταυτικές ροές έχουν ε, μειωθεί Και επίσης και το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στο πλευρό σας παρά το Brexit. Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη και αν μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο στο αποτέλεσμα, στο να μας το πείτε. Ο Ιβο Βάγκο, εισηγητής για το θέμα της Μακεδονία από το Άλντε. Συγχαρητήρια. για την διαπραγματευτική σας τακτική και στους δύο πρωθυπουργούς της ε, χώρας και της ε, Ελλάδας. Κάνατε εξαιρετική δουλειά σε κάτι που για πολύ καιρό φαινόταν αδύνατο. Έχετε λοιπόν ε, δώσει ένα νέο πρότυπο για το πώς μπορούν να ενισχύσει τα Βαλκάνια. Θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα, το δημοψήφισμα θα πρέπει να αποτελέσει γεγονός που θα ενώσει τους πολίτες της, Μακεδονίας. Ε, όλα τα κόμματα θα πρέπει να ε, τηρήσουν τις δεσμεύσει της Συμφωνίας του Πριζίνο. Τα κόμματα θα πρέπει να θέσουν ε, σε πρώτη σειρά το συμφέρον της χώρας και όχι να υποφεληθούν ε, πολιτικά. Πώς λοιπόν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξει ενότητα όσον αφορά αυτό το σημαντικό ερώτημα για την Μακεδονία. Πώς θα συνεργαστείτε με την αντιπολίτευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ήβο για τους πράσινους τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε ξανά. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Είμαστε οι πιο σύλληψεις προς την ε, υποστήριξη της ε, ένταξης της χώρας σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θέλω να συγχαρώ, να συγχαρώ για την ιστορική διπλωματική ε, νίκη και ελπίζω να στεφθεί και με ένα πετυχημένο δημοψήφισμα. Το ερώτημά μου δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά με ένα θέμα που έχει να κάνει με μεταρρυθμίσει. Κάνετε λόγο για ανάγκη να υπάρχει ανταγωνισμό στι μεταρρυθμίσει στην περιοχή. Κάτι το οποίο προσυπογράφω. Υπάρχει όμω ένα τομέα στον οποίο χρειάζεται συντοσμό και τοπική περιφερειακή συνεργασία και αυτό είναι η καταπολέμηση τη διαφθορά. Μπορεί να δώσει νέα όθηση η κυβέρνησή σα στην ήδη ε, συνεργασία και τα μέτρα για την ε, καταπολέμηση τη διαφθοράς. Ευχαριστώ, Τόμας. Για την ΚΟΕ θα δώσω το λόγο τώρα στον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Παπαδημούλη. Κύριε Δημητρόφ, σας καλωσορίζω στην συνεδρίασή μας και θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά και σας και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, για την ιστορικής σημασίας συμφωνία που συνυπογράψατε και την οποία, όπως διαπιστώνετε, χαιρετίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ότι στο δημοψήφισμα που θα οργανωθεί σε ένα περίπου μήνα στη χώρα σας, αυτή η συμφωνία θα εγκριθεί από το λαό σας και έτσι η χώρα σας θα ονομάζεται από τούδε και στο εξής Βόρεια Μακεδονία, λύνοντας με έναν κοινά αποδεκτό τρόπο μια διαμάχη που ταλαιπώρησε τους λαούς μας και τις χώρες μας για πολλές δεκαετίες. Σημειώνω με ικανοποίηση την ε, δέσμευσή σας ως κυβέρνηση να προωθήσετε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, την καταπολέμηση της διαφθοράς και το σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας σας, όπως και όλων των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση και το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουν ολόθερμα τη συμφωνία και περιμένουν την, ε, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στα δικά μας βήματα. Το ερώτημά μου είναι αν υπάρχουν χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά τη γνώμη σας εργάζονται για να μην υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. E Ευχαριστώ για το EFTD, ο κύριος Κασάλντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω. Αυτό ο οίκος είναι και δικό σας οίκος και οίκος του λαού σας. Είναι ιστορικό γεγονός το οποίο στο οποίο ενδιαφερόμαστε σήμερα και είναι σημαντικό να συγχαρούμε και εσάς και τους Έλληνες φίλους για αυτή την ιστορική συμφωνία και να σας χαρούμε και για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθείτε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την εκστρατεία που γίνεται για το προσεχές δημοψήφισμα. Θα κάνετε έναν εθνικό διάλογο στον οποίο θα συμπεριλάβετε την κοινωνία των πολιτών, τους ακαδημαϊκούς ε, και τα μέσα μας ενημέρωσης για να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σημασία του και να ε, αντικρούσετε τα κόμματα που θέλουν να μποϊκοτάρουν την προσπάθειά σας. Σύντομα θα βρεθώ στα Σκόπια για να ασχοληθώ με τη συμμετοχή της νεολαίας στην πολιτική. Άρα, η συμμετοχή της νεολαίας είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ποιο είναι το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ε, για να προσέλθει η χώρα σας στο ΝΑΤΟ. Και όσον αφορά το θετικό ανταγωνισμό, θεωρώ ότι η χώρα σας θα μπορέσει να αποτελέσει ένα φωτεινό παράδειγμα για όλη την περιοχή. Άλλες διερωτήσεις θα κάνουμε τον πρώτο γύρο απαντήσεων και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, για να δώσουμε και ένα ρωμαλινικό, Ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δημητρόφ, σας καλωσορίζω. Μιλήσατε με συνένεση και οριμότητα. Όμως να σας κάνω ένα ερώτημα. Ρώτησα ένα κάτοικο της Νέας Υόρκης και ένα κάτοικο της Νέας Ζηλανδίας. Πώς ονομάζονται, πώς αυτοπροσδιορίζονται. Και μου απάντησαν Νεοϊορκέζος και Νεοζηλανδός. Με τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου στις Πρέσπες μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης των Σκοπίων. Το κράτος θα ονομάζεται Βόρειος Μακεδονία. Εσείς πώς θα ονομάζεστε. Βορειομακεδόνας ή Μακεδόνας. Γιατί αν ονομάζεται Μακεδόνας, πρέπει να μας εξηγήσετε αν η εθνότητα που ζει σήμερα στην περιοχή της Σφύρομ ήρθε τον 6ο μετά Χριστό αιώνα στην περιοχή, πώς γίνεται να ονομάζεστε Μακεδόνες. Εάν το θέμα με τη Μακεδονία ξεκίνησε από την τρίτη κομμουνιστική διεθνή, γιατί ο Στάλιν είχε κάποιες βλέψεις στο Αιγαίο εκείνη την εποχή, ή από τον Τίτο στα τέλη της του 1940 που δημιούργησε μακεδονική εθνότητα, μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εκκλησία, γιατί αυτό πρέπει να είναι κομμάτι της συμφωνίας. Το κόμμα μου, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια συμφωνία. Πώς νομιμοποιεί δύο έννοιες, οι οποίες δημιουργήθηκαν την εποχή του Τίτο, μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά στην Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης και εσείς ε, Έλληνας από την Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, ε, τότε είναι γεμάτη η αίθουσα σήμερα. Φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον να ενταχθούν και η δική σας χώρα, αλλά και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσωπικά ως Έλληνας είναι ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, διότι θέλω να υπάρχει μια λύση στο ονοματοδοτικό, στο θέμα της ονομασίας, αρκεί να είναι μια λύση εθνικά αξιοπρεπή για του δύο λαού, με σεβασμό στην πραγματική ιστορία, χωρί τι καπηλίε, τη ιστορικέ που ζήσαμε στο παρελθόν. Έχω λοιπόν να σα κάνω ένα σαφέστατο ερώτημα. Εάν, επειδή το ερώτημα του δημοψηφίσματο δεν είναι ναι ή όχι συμφωνία, αλλά είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη, ο λαό ψηφίσει ναι στην είσοδο στην Ευρώπη. Αλλά μετά από λίγο καιρό, η εκφρασμένη βούληση του λαού στο κοινοβούλιο σα, δεν βρει μια πλειοψηφία συνταγματική αναθεώρησης, κοινώ η κυβέρνησή σα δεν βρει 81 βουλευτέ στου 120 για να προχωρήσει στι συνταγματικέ αλλαγές που έχετε συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση. Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα γίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών. Αν λοιπόν ο λαό πει ναι στο δημοψήφισμα, αλλά δεν βρεθούν οι 81 στου 120 βουλευτέ για να προχωρήσει η συμφωνία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τον πρώτο γύρο. Μπορείτε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, ε, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά περίπου, μέχρι τις 10 και 4. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ευγενικά σας λόγια, για τις καλές ερωτήσεις και για τις δύσκολες ερωτήσεις. οι σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων. Εγώ δεν θυμάμαι μία περίοδο χρονικά που να είχαμε πιο χαλαρές ε, σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων στη χώρα. Η κρίση εισήγαγε ένα νέο στοιχείο στις σχέσεις μεταξύ των μακεδονικού λαού και των άλλων εθνοτικών ε, κοινοτήτων, γιατί υπήρχε να αναγνώριση ότι είμαστε στην ίδια βάρκα, στην ίδια κατάσταση και ιδίως κέντρα. Ξαφνικά συνειδητοποίησαν οι άνθρωποι ότι όλοι είναι κατά της διαφθοράς, ότι όλοι θέλουν λογοδοσία και δικαιοσύνη και αυτό δημιουργεί μια πρόκληση στο σημερινό πολιτικό τοπίο στη χώρα. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εθνικό. Η εθνική ε, ατζέντα, στρατηγική, ε, μπορεί να μην αρκούν σε ορισμένες περιπτώσεις. Όταν οι χώρες προδεύουν, τότε διαδίδεται η ελπίδα στις ε, κοινωνίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παράγοντα. Τώρα περιμένουμε κι εμεί να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε το δημοψήφισμα και μια συνταγματική διαδικασία. Στο μέλλον έχουμε ξεκινήσει τι συνομιλίε με τον ΝΑΤΟ για την προσχώρηση και ανυπομονούμε να ξεκινήσουν και διαπραγματευτικές συνομιλίες ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρηση. Και έχουμε μια σταθερή πολιτική, μια κοινωνία για όλους. Είναι πυλώνας της κυβέρνησης αυτής. Κάποιες ερωτήσεις αναφέρθηκαν σε ελοδοπή παρέμβαση. Υπάρχουν δυνάμεις που δεν είναι ικανοποιημένες όταν βλέπουν την επίλυση των προβλημάτων και την επίτευξη πρόοδου για μας, κυρίως για το θέμα του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι εδώ το ΝΑΤΟ είναι ένας μεγάλος συντελεστής. Στην εξίσωση για μας ε, είναι κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί. Μία ιστορική αποστολή που δεν έχει ολοκληρωθεί. Την ξεκινήσαμε το 1993 όταν το κοινοβουλίο μας ομόφωνα αποφάσισε ότι θέλουμε να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η αποφασή μας. Η κοινή γνώμη συνεχώς ε, ε, κατά τα 2, 3, 3, 4 υποστηρίζει αυτό το στρατηγικό στόχο και έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα στην περιοχή μας. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε πολιτικούς ανταγωνισμούς δια Και πιστεύω ότι οι δυνάμεις αυτές θα συνειδητοποιήσουν ότι αν επιληθούν τα ζητήματα ε, και προ προοδεύουν και τα Βαλκάνια, είναι καλό και για αυτέ τι δυνάμει. Ίσως να μην έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά θα καταλήξουμε εκεί μακροπρόθεσμα. Επαγρυπνούμε, βάζουμε τα δυνατά μα, ε, έχουμε βοήθεια από φίλους και συμμάχου για να διασφαλίσουμε ότι ενημερώνονται οι πολίτε γιατί αν δεν ενημερώνονται οι πολίτε, αποτυγχάνει η δημοκρατία. Μπορούν να κάνουν τι σωστέ αποφάσει μόνο όταν είναι ενημερωμένοι. Το κάνουμε αυτό λοιπόν, αλλά δεν είναι εύκολο και έχουμε και το δημοψήφισμα και εσείς ε, στην Ευρώπη έχετε και σχετική εμπειρία με δημοψηφίσματα. Έτσι λοιπόν βάζουμε τα δυνατά μας ε, για να έχουμε την ορθή απεύθυνση στους πολίτες, να τους ε, ενημερώσουμε και να είναι ελεύθεροι να λάβουν τις αποφάσεις για το μέλλον τους. Τώρα πώς θα δημιουργήσουμε πολιτική ενότητα στο εσωτερικό. Είχαμε την ερώτηση από τον κύριο Ιβο Βάγκλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα το μαθαίνουμε. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να συνεργαστούμε στο να διατυπώσουμε την ερώτηση. Υπήρξαν πολλοί πολιτικοί συμβασμοί και για τη σύνθεση της Εκλογικής Επιτροπής, για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, είχαμε νέους κανόνες. Δεν ε, έχουμε καταλήξει ακόμη. Στο αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσε ότι δημοσίως θα ενημερώσουν ε, το κοινό για τη θέση τους ε, σχετικά με το δημοψήφισμα στις αρχές Σεπτεμβρίου, γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου. Αν ε, θέλω να είμαι κακός, αυτό μου υπενθυμίζει το μικρό μου γιο που θα είναι 5 το Σεπτέμβριο και το ρωτάω γιατί έχει θυμώσει και μου λέει δεν θα σου πω σήμερα, θα σου πω αύριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Ακούσαμε και τη φράση του big to fail» ε, με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση το 2010. Είναι ιστορική αυτή η διαδικασία. Δεν ε, πρόκειται για μένα, ούτε για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ζαεφ, ούτε περί κυβέρνησης υπερπολιτικών κομμάτων πρόκειται. Πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία να κλείσουμε ένα δύσκολο ζήτημα και να ανοίξουμε την πόρτα για το μέλλον. Πρέπει να υπάρξει πολιτικό φύγημα για την αντιπολίτευση όχι να κατασταθεί πιο δύσκολη αυτή η διαδικασία, να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη και κατόπιν να επιτεθεί στην κυβέρνηση, όπως ε, κάνουν συνήθως για την οικονομία, για διάφορα θέματα, αλλά όχι για αυτό το ζήτημα. Σε αυτή την διαδικασία ορίμανσης ε, και για την χώρα μας, αλλά και για την περιφέρεια, έχουμε τις προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και εμείς, αλλά και αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν αυτή την ιστορική ευθύνη. Και αυτό δεν μπορεί να σχετιστεί με τη λογοδοσία για την επίθεση στο Κοινοβούλιο, ούτε με την λογοδοσία σε σχέση με τους ισχυρισμούς του 2015. Αν ε, θέλεις να είσαι μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, θα πρέπει να σέβεσαι κάποιες αρχές, κράτος δικαίου και λογοδοσία. Δεν μιλάμε εδώ για πολιτικές ιδεολογίες. Δεν πρόκειται περί πολιτικών ιδεολογιών. Τώρα, η καταπολέμηση της διαφθοράς στην περιοχή νομίζω είναι κάτι απαραίτητο. Υπάρχουν δύο μεγάλα δεινά στα Βαλκάνια, οι πελατικές σχέσεις και η διαφθορά. Θα πρέπει να τα καταπολεμήσουμε και τα δύο είναι πιο εύκολο να τα καταπολεμήσουμε όταν ε, συμμετέχουμε στην ε, διαδικασία προσχώρησης, γιατί η διαδικασία αυτή είναι ο καλύτερος ε, τρόπος καταπολέμησης αυτών των φαινομένων. Ξεκινήσαμε τη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου δημόσιων εισαγγελέων για να συνεργαστούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, γιατί η ερώτηση αφορούσε την διασυνορική συνεργασία, την περιφερειακή συνεργασία στο θέμα αυτό. Τώρα για την εκστρατεία που ξεκινάει αύριο θα είναι πράγματι πολύ ευρεία, γιατί θα συμμετέχουν μόνο τα πολιτικά κόμματα, αλλά και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα συμμετάσχουν. Κάθε πέμπτη ε, μπαίνω στο facebook και απαντώ στις ερωτήσεις ε, που μου στέλνουν οι πολίτες καθ' όλη την εβδομάδα για τη συμφωνία, διάφορα άρθρα της συμφωνίας γιατί συμφωνήσαμε στο ένα γιατί δεν ε, συμπεριλαμβάνεται κάτι άλλο και θα συνεχίσουν να το κάνω αυτό. Τώρα για τον είμαι Μακεδόνας, είμαι Μακεδόνας. Μου θέσατε αυτή την ερώτηση. Όταν η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, θα λέγεται η χώρα μου Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, θα είμαστε Μακεδονές που θα μιλούν τη μακεδονική γλώσσα, αναγνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα όρος Μακεδόνας έχει διαφορετικές σημασίες. Και στην Ελλάδα υπάρχουν Μακεδόνες και δεν ε, θα μπω τώρα σε έναν ορισμό για το πώς προέκυψε ε, με όρους ε, αρχαίας ιστορίας, η περιφερειακή κληρονομιάς, αλλά το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στον αυτοπροσδιορισμό στην Ευρώπη το 2018, τον 21ο αιώνα, είναι κάτι αναμφισβήτητο. Η συμφωνία αυτή βασίζεται σε δύο πυλώνες. Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ της χώρας Μακεδονίας και της περιοχής Μακεδονίας στην Ελλάδα. Η διάκριση αυτή είναι έργα για κάθε σκοπό θα πρέπει να περάσουμε τη δύσκολη διαδικασία του να αλλάξουμε το Σύνταγμά μας, γιατί θέλει ο γειτονάς μας να το πράξουμε και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δύο ευρωπαϊκές χώρες που είναι γείτονε θα πρέπει να μπορούν να δεκτούν η μία την άλλη και για το πώς νιώθουν οι πολιτικοί δεν μπορούν να αλλάξουν τις ταυτότητες. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι αποτέλεσμα μιας ιστορικής διαδικασίας και δεν μπορούμε να το αγγίξουμε αυτό, να το θίξουμε αυτό. Και γι' αυτό αναφέρομαι στη διαδικασία αυτή σαν μια διαδικασία ενηλικίωσης και αν ε, το κάνουμε σωστά, αν ε, έχουμε επαρκή φιλία και γνωριστούμε καλύτερα, σε πέντε χρόνια, στο 2023, θα βλέπουμε το παρελθόν και θα αναρωτιόμαστε πώς ε, είναι δυνατόν να μην έγινε αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 90. Χάσαμε τόσο πολύ χρόνο, χάσαμε μία γενιά. Θα μπορούσαμε να ήμασταν και τότε φίλοι, θα είμαστε τώρα φίλοι και στο μέλλον. Και θα ηρεμήσει η κατάσταση. Θα σταματήσω εδώ γιατί αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Second round Ευχαριστώ. Ας περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Η κυρία Σακοράφα, και όντως η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Υπουργό στην Επιτροπή μας. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως. Γνωρίζουμε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα τεράστια συμφέροντα και οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί που χαρακτηρίζουν τη σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση στην περιοχή. Οι διαφωνίε μου με του σχεδιασμού αυτού είναι πολιτικέ, έχουν αναφερθεί πάρα πολλέ φορέ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, αλλά και όπου αλλού μου δόθηκε η ευκαιρία. Σας ρωτώ λοιπόν, αν πιστεύετε ότι αυτή η ολοκληρωτική και ουσιαστικά ανεφόρον πρόσδεση της κυβέρνησης και του κράτους σας με αυτά τα συγκεκριμένα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα προς όφελο του λαού σας με δεδομένο και όλα στο βίο παρελθόν της περιοχής και την δημιουργία όλων αυτών των κρατών στη συγκεκριμένη περιοχή. Σας ευχαριστώ. Thank you, dear colleague. Ευχαριστούμε, συνάδελφα. Κυρία Σουίτσα. Thank you, David. Ευχαριστώ, David. Θα μιλήσω τη μητρική μου, εφόσον και αυτή είναι σλαβική γλώσσα. Λοιπόν, ε, δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τους γειτονές του, την οικογένειά του, αδιαφυσβήτητα. Αυτό είναι μια καλή αφετηρία είπατε ότι η περιοχή αυτή δεν είναι νησί, ούτε η Μακεδονία, απλώς ε, περιστοιχίζεται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα εναπόκειται σε μία γενιά να αναλάβει αυτό το ιστορικό καθήκον και προφανώς η δική σας γενιά είναι αυτή που θα πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Μιλήσατε για μια διαδικασία ενηλικίωσης, ακριβώς ε, αυτό είναι. Όλοι πρέπει να μάθουμε πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Και αυτή η ειρήνη που απολαμβάνουμε τώρα στην περιοχή και εμείς, η Κροατία που είμαστε στην ε, ευρύτερη περιοχή, εκεί βρισκόμαστε. Ε, βέβαια δεν θέλουμε να την αποκαλούμε Βαλκάνια, Νότια νότιο-ανατολική Ευρώπη. Είναι σίγουρα το μεγαλύτερο επίτευγμα των ε, τελευταίων ετών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να πετύχετε συνένεση με την αντιπολίτευση, γιατί μόνο αν υπάρχει αυτή η ενότητα στο εσωτερικό της χώρας θα είναι πιο εύκολο να λειτουργήσετε καλύτερα στις σχέσεις σας με τις γειτονικές χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σίγουρα είναι μία από τις απαιτήσει με βάση τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καϊλή. από τους σοσιαλιστές, παρότι κάθεται στα έδρανα του ΕΛΚ. Ναι, είμαι επισκέπτρια εδώ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τον, για λόγο. Καλώς ήρθατε. χαίρομαι που οι γειτονές μας έχουν διάθεση διαλλακτική από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ε, και την πρόθεση φυσικά να ξεπεράσουν χαρακτηρισμούς αλυτρωτικούς αλλά και μια ρητορική που θα συμφωνήσω επί πολλά χρόνια πλήγωνε τις σχέσεις μας. Επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ τυχεροί που η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει δείξει αυτή τη ε, διάθεση μετά από πολλά χρόνια. Ε, Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και οικονομικές σχέσεις οι λαοί ε, συνέχιζαν να συνεργάζονται σε πάρα πολλά επίπεδα. Το γνωρίζετε, έχουμε επισκεφτεί τη χώρα σας και, φυσικά πάρα πολλοί επισκέπτονται την Ελλάδα διαρκώς. επιτρέψτε μου όμως να ρωτήσω αν αισθάνεστε πως απαιτείται να διορθωθεί η συμφωνία μέχρι την ολοκλήρωσή της καθώς θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου ότι υπάρχει το παράδοξο να είναι η ονομασία Βόρεια Μακεδονία, αλλά η στρέβλωση να μην διευκρινίζει ότι αυτό θα είναι και το, ο προσδιορισμός των κατοίκων. Καθώς σας είπα, ε, εγώ από τη Μακεδονία θα πρέπει να εξηγώ ότι οι κυβερνήσεις μας δεν διόρθωσαν να, ε, ή παρέλειψαν να διορθώσουν αυτό το παράδοξο. Επίσης, αναφέρατε ότι οι γείτονε ε, ζητούν επιληθεί και το ΝΑΤΟ ως ε, chair του ΝΑΤΟ εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο το ΝΑΤΟ δεν θέλει να εσωτερικεύσει τέτοιε διενέξει, οπότε θα είναι υποαίρεση η συμφωνία αν δεν γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και να ρωτήσω και ένα τελευταίο, αν υπάρχει και μια ειδική επιτροπή που θα λύσει και ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν οικονομικά, για παράδειγμα κάθε προϊόν που ονομάζεται μακεδονικό ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστούμε την Εύα Καϊλή. Ο κύριος Χιτζουκ από την Άλντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα διπλωματικά σας επιτεύγματα. Εδώ βρίσκομαι. Φυσικά εδώ πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και επικριτική αλλά και βοηθητική. Ένα ερώτημα λοιπόν προς εσάς είναι πώς εμείς ως Ευρώπη μπορούμε να σας βοηθήσουμε για την επιτυχή έκβαση του δημοψηφίσματος. Και βέβαια σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το δημοψήφισμα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πέτρελ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα πολύ θετικά λόγια που εκφράσατε υπέρ της Ευρώπης. Πιστεύω ότι η χώρα σας έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική, καθώς και ολόκληρος ο Νότος, ολόκληρη η περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εγώ είμαι μέλος ε, της κοινή Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ε, θα συνεδριάσουμε σύντομα στα Σκόπια Χαίρομαι που πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή τώρα μπορεί να συνεχίσει το έργο της. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή τη διαδικασία και ελπίζω οι πολιτικές εξελίξεις να ακολουθήσουν την φιλοευρωπαϊκή άγουσα. Ελπίζω να μην υπάρχουν άλλα τέτοια ζητήματα για την απειλή της ε, ταυτότητά σας. Παρακαλώ. Um, chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε και σε χαρητήρια για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να πω ότι παρότι εύχομαι καλή επιτυχία για τον μέλλον των προσπαθειών της χώρας σας, παρόλα αυτά τα δημοψηφίσματα είναι απρόβλεπτα πράγματα. Και για στον Βασίλειο το γευτήκαμε κανονικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ποια είναι η προετοιμασία που κάνετε σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα. Θα γίνουν ε, κοινοβουλευτικές εκλογές. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ήδη ακούστηκε το ζήτημα του μποϊκοτάζ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τίθεται λοιπόν τέτοιο θέμα Ήθελα απλώ να πω ότι είναι δύσκολο το θέμα του δημοψηφίσματο. Γενικά να το ξέρετε ότι είναι κάτι το απρόβλεπτο. Κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη παρατήρηση θέλω να κάνω. Αφού έχω συναντήσει πολλούς υπουργούς εξωτερικών από τα Σκόπια, καταρχάς να σας συγχαρώ για τη συμφωνία είναι κάτι για το οποίο πρέπει να χαιρόμαστε και να σημειώσουμε ότι θα πρέπει όλοι οι δυνάμεις στη χώρα σας να στηρίξουν αυτή την λύση, γιατί είναι μια ιστορική ευκαιρία που δεν θα πρέπει να προσπεράσετε. Και τρίτον, είναι μια καλή ένδειξη και για το αντίστοιχο κόμμα με το δικό μου στη χώρα σας. Δηλαδή ότι όλοι στη χώρα σας και οι μειονότητες όπως είναι οι Αλβανοί θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Ε, και αυτό θα γίνει μόνο αν εγγυηθεί η ασφάλεια και σταθερότητα στη χώρα. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. von Ballen. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Επικροτώ τα όσα είπε ο κύριος Μπροκ για την στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων για την συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζοφκό, τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, αλλά δεν το είχαμε σημειώσει αυτό το όνομα. Έχουμε και άλλους ομελετές, λοιπόν. Ηρεμία. Εγώ μπορώ να δώσω μόνο το λόγο σε όσους έχουν καταγραφεί στον κατάλογο. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Πετικόβε, Κόβετσεφ, Κέλλα. Υπάρχει κάποιος άλλος. Όχι. Ωραία, κυρία Ζόφκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό Δημητρόφ. Συμφωνώ και με τους υπόλοιπους συναδέλφους και εγώ προέρχομαι από αυτή την ε, ευρύτερη περιοχή. Ξέρω την αξία της ε, ειρήνης και της σταθερότητας Επομένω, στηρίζω πλήρω τι προσπάθειέ σα ε, για να εξευρεθεί μια κοινή λύση και με την αντιπολίτευση και με όλε τι μειονότητε, όπω είπε και ο κύριο Μπροκ. Ε, ναι, πρέπει να υπάρχει και μια στρατηγική επικοινωνίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την ταυτότητα. Και εγώ το γνωρίζω αυτό γιατί για πολύ καιρό μοιραζόμαστε την ίδια επικράτεια, αλλά από πλευρά μα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμεί για να μεταφέρετε καλύτερα αυτό το μήνυμα τη ε, ειρήνη και σταθερότητα στα Βαλκάνια. Να έχουμε μια ειρηνική λοιπόν Μακεδονία που θα εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το σημαντικό και έχετε φίλου εδώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπιτικόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και εγώ συμμετέχω στην ομάδα φίλη της Μακεδονίας του Κοινοβούλιο. Σήμερα όμως κατά βάση θέλω να επικροτήσω και να εκφράσω το θαυμασμό μου για το πολιτικό σας θάρρος και την πολιτική λογική ε, που επικράτησε και στις δύο πλευρές, και στα Σκόπια και στην Αθήνα, για να εξευρεθεί αυτή η λύση. Ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις μόνο. Πρώτον, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρξει τρόπος και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να έχουν ένα θετικό αφήγημα για την λύση αυτή. Και δεύτερον, είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ε, να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα εάν ε, είμαστε αμετακίνητοι στην προσήλωση και στην αποφασιστικότητά μας και να είμαστε ξεκάθαροι ότι θέλουμε τη Μακεδονία, την δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας των μέλλον, να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διστάσουμε να ξεκινήσουμε την ενταξιακή διαδικασία. Ευχαριστώ. Άντρη Ευχαριστώ πολύ, Ντέιβιντ. κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το θάρρος σας και τη δύναμη που επιδείξετε για να φέρετε τη Μακεδονία στον ε, χώρο της συνταξιακής διαδικασίας μετά από τόσα χρόνια ανεπίλητων διαφορών. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Έχει Έχουμε υπογράψει και συμφωνία μεταξύ μας. Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τους ε, Μακεδόνες γείτονες και φίλους ε, για να ακολουθήσουν την ενταξική διαδικασία των συμμετρών δυνατών. Υπάρχουν κάποια λεπτά ζητήματα που εθίγησαν προηγουμένως και εσείς ε, επισημάνατε ότι ο αυτοπροσδιορισμός και η ταυτότητα είναι μία ιστορική διαδικασία ε, μιλήσατε και για την Επιτροπή Κάρνεγκη. Ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε σωστά πράγματα, αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Εάν ένας Μακεδόνας θεωρεί ότι είναι Μακεδόνας, μπορεί να λέει ότι είναι Μακεδόνας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει την ταυτότητα κάποιου άλλου ή και την ταυτότητα των θανόντων. Ήταν αυτοί που ήταν. Τώρα αν ήταν ναι, μια δικατορία, ο Τίτο, δεν ξέρω ποιος, όποιος και να ήταν, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει ε, την ταυτότητα των νεκρών. Σα εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στον ευρωπαϊκό δρόμο που θα ακολουθήσει η ε, Δημοκρατία της Μακεδονίας και εσείς προσωπικά. Ευχαριστώ τέλο ε, τον Ανικέλα. Ευχαριστώ πολύ, Ντέιβιντ. Κύριε Υπουργέ. Συμφωνούμε απολύτω ότι είναι κοινά τα συμφέροντα και κοινό το μέλλον. Γιατί χρειαζόμαστε και εμείς τη Μακεδονία ω πλήρε μέλο ακριβώς όπως χρειάζεται και η Μακεδονία την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν, αλλά μπορούν να γίνουν και ε, κατά τη διάρκεια της επίσημης πρωταξιακή διαδικασίας. Ένα ερώτημα τώρα. Μας προβληματίζει όλο ένα και περισσότερο εδώ η αυξανόμενη ρωσική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια. Ιδίως ε, σε ό,τι αφορά την ρωσική αντίθεση στην ένταξή σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Την ένταξη των χωρών των Βαλκανίων, όπω ε, στο Μαυροβούνι για παράδειγμα. Υπήρξαν περιπτώσει ε, στήριξη και χρηματοδότηση από τη Ρωσία εκστρατιών παραπληροφόρησης ε, στη Μακεδονία και στην Ελλάδα υπήρξαν ανησυχητικά φαινόμενα. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Πρόσφατα ορίστηκε μία εκλογική επιτροπή. Θεωρείτε ότι θα διευκρινιστούν εκλογικοί κατάλογοι με ικανοποιητικό τρόπο πριν από το δημοψήφισμα. Ωραία. Ελπίζω να πήραν το λόγο όσοι ήθελαν. Νίκολα, Έχεις 10 λεπτά για να απαντήσεις όσο γίνεται σε περισσότερα ερωτήματα. Thanks, David. I'll... Στο David θα προσπαθήσω. Υπήρξαν πολλά θετικά σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιες ερωτήσεις για την αντιπολίτευση και ανησυχίες εκφράστηκαν και είναι δικαιολογημένες και για να είμαι δίκαιος Έχουμε διαφορετικές φωνές από εκείνη την πολιτική, από εκείνο το πολιτικό στρατόπεδο. Κάποιες τονίζουν την ευθύνη της αντιπολίτευσης, τη δικιά τους ευθύνη όσον αφορά τη συμφωνία, το μέλλον, το δημοψήφισμα. Κάποιες είναι ακόμα και υπέρ της συμφωνίας, ε, δεν το λένε ξεκάθαρα, αλλά είναι προφανές στα μέσα μας ενημέρωση. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει ένας λόγος να είμαστε αισιόδοξοι, αν και όταν ο αρχηγός κάνει λόγο για τη συμφωνία, αναφέρει ότι είναι παράδοση άνευ ε, είναι λεγόμενη, ε, αναφέρεται σε αυτήν ως λεγόμενη συμφωνία και κάνει λόγο για παράδοση. Είναι δύσκολο λοιπόν για εμένα που δεν συμμετέχω σε κάποιο πολιτικό κόμμα κατά τύχη πολιτικός θα έλεγα ότι είμαι δεν θεωρώ τον εαυτό μου εμπειρογνώμονα έχω υποστηρικτές έχω δώσει υποσχέσεις και για μένα είναι αδιανόητο σε μια στιγμή σαν κι αυτή να μην σκεφτόμαστε τη χώρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το δικό μου πολιτικό μέλλον και το γνωρίζω και για τον Πρωθυπουργό μας. Είναι πολύ πιο σημαντικό το ζήτημα. Αν το κάνουμε σωστά, η χώρα θα πορευθεί σωστά και θα είμαστε όλοι καλύτερα. Τα κόμματα αλλάζουν, είναι στην αντιπολίτευση, στην κυβέρνηση. Όμως αυτές τις ιστορικές στιγμές πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Έκανα επαφές ε, με φίλους Έλληνες στο πλαίσιο αυτό και τώρα τον που θέσετε για το κοινοβούλιο υπάρχουν τρία κίνητρα για αυτή τη συμφωνία. Το ένα είναι να χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας με τους γειτονικού λαούς το δεύτερο είναι να ξεκλειδώσουμε την πόρτα για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, για, την, διαπραγματεύσεις και για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και εμείς και οι φίλοι μας οι Έλληνες θα είμαστε καλύτερα αν το πετύχουμε αυτό. Πιστέψτε με, για κάποιους στη χώρα μου είμαι ήρωας, για άλλους είμαι προδότης και ο Νίκος είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς στην Ελλάδα. Αν θα μπορούσα να γράψω τη συμφωνία μόνος μου θα ήταν μια καλύτερη συμφωνία από τη δικιά μου την οπτική. Αν ο Νίκο είχε το δίκαιο να γράψει μόνο του, να τη συντάξει μόνο του τη συμφωνία, θα ήταν μια καλύτερη συμφωνία από την ελληνική οπτική. Το γεγονό ότι έπρεπε να την συγγράψουμε και να συμβαστούμε και να προστατέψουμε ό,τι είναι πιο σημαντικό ε, για την Ελλάδα και αντίστοιχα για την ε, δική μου χώρα, αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί αυτή είναι η έννοια του συμβασμού αν σκεφτόμασταν μόνο πώς θα το εκλάβουν τώρα αυτό στην Αθήνα ή στα Σκόπια, δεν θα το είχαμε υπογράψει ποτέ το κείμενο. Αλλά σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια από τώρα, τα ωφέλη θα είναι τόσο μεγαλύτερα που θα κοιτάμε πίσω και θα αναρωτιόμαστε πραγματικά γιατί δεν το κάναμε αυτό 20 χρόνια νωρίτερα. Μπορεί κανείς να βιοποριστεί ως πολιτικός μέσω των διαμαχών ή να επιλύσει τις διαμάχες και να δώσει ζωή, σταθερότητα στους ε, πολίτες και στους φυσικούς σύμμαχους. Ε, τέθηκε ερώτημα για την ιστορία. Θεωρώ ότι σήμερα στην Ευρώπη και ειδικά σε μια για την οποία ο Ούσαν είπε ότι παράγει υπερβολική ιστορία, την οποία δεν μπορεί να χωνέψει. Όλες οι χώρες έχουν τα ιστορικά τους αφηγήματα. Και όλες οι χώρες είναι περήφανες. Δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό που μπορούμε να πετύχουμε σήμερα. Να δημιουργήσουμε αυτοκινητόδρομους προς τη Βουλγαρία και να αυξήσουμε το εμπόριο, να το διπλασιάσουμε. Όταν όμω κάνουμε λόγο για έθνη, πώς θα αισθανόσασταν αν ο γείτονα σας έλεγε ότι το έθνος σου είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα. Όλα τα έθνη είναι τεχνικά κατασκευάσματα. Και στη φιλοσοφική σκόψη είναι κατηγορία του 18ου και του 19ου αιώνα. Και όλα στηρίζονται από ένα αφήγημα. Το κλειδί εδώ είναι τα ιστορικά μας αφηγήματα να μην είναι ενάντια στους γειτονέ μας, αλλά να τους συμπεριλαμβάνουν. Και αυτή είναι μια διαδικασία την οποία, από την οποία πέρασε και η Γαλλία και η Γερμανία και χρειάστηκαν δεκαετίες. Μην ε, αναμένετε λοιπόν αποτελέσματα σε μια νύχτα. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα και θα φτάσουμε και στο στόχο μας. Θεωρώ ότι το σημαντικό είναι να εστιάζουμε στο σήμερα και στο αύριο και να αφήσουμε τα υπόλοιπα στους ε, ιστορικούς. Εγώ είμαι νομικός, έχω σπουδάσει διεθνές δίκαιο. Αν θα επιτύχει η συμφωνία, αν το Σύνταγμα θα αλλάξει, ε, το δημοσίευμα δεν είναι ε, νομοθετική προπόθεση για τη συμφωνία. Κάνει λόγο η δυνατότητα δημοψήφισματο η συμφωνία. Ο λόγο που το κάνουμε όμω το δημοψήφισμα είναι πρώτον ότι έγινε έγιναν το λόγο του πολιτικού διαλόγου τελευταία χρόνια. Το επιθυμούν όλα τα πολιτικά κόμματα. Και για να εφαρμόσουμε την ε, συμφωνία, χρειαζόμαστε δύο τρίτα της πλειοψηφία ε, στην Βουλή για την ε, σταγματική μεταρρύθμιση. Αν μα στηρίξει ο κόσμο, αν κερδίσουμε τον κόσμο με το μέρος μας, τότε θα είναι δύσκολο οποιοδήποτε στο Κοινοβούλιο να πει όχι και θα πετύχουμε την πλειοψηφία των δύο τρίτων. Όσον αφορά τις ε, παρεμβολές στο εξωτερικό, ως υπουργό Εξωτερικών δεν είναι σοφό από την πλευρά μου να αναφερθώ σε λεπτομέρειες και να μιλήσω για τους φίλους μας, τους Ρώσους, δημοσίω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρώτον, ε, όσον αφορά το σήμερα, το αναλαμβάνουμε σαν δικιά μας προσωπική ευθύνη χωρίς ξένες παρεμβολές. Όμως κάποια στιγμή όλοι θα καταλάβουμε ότι μια σταθερή σταθερότητα στην περιφέρεια, στην περιοχή είναι προς δικός μας όφελος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους Ρώσους. Δεν βλέπω άλλο τρόπο για το μέλλον, για να μην υπάρχει ένταση μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πώς θα το πετύχουμε να έχουμε μια αξιόπιστη δικαστία, αξιόπιστη δικασία προσχώρησης και με το να προσεγγίσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει να κάνει με καθημερινή πολιτική, αλλά ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης να εξάρουμε όταν έχουμε τις επιτυχίες. Αυτές είναι τρεις γραμμές στις οποίες μπορείτε να μας βοηθήσετε. Το βασικό είναι να τηρήσουμε τη Συμφωνία της Ελληνικής του 2003. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Βαλκάνια, έχουμε αντλήσει διδάγματα, είναι πολύ πλοκή η διαδικασία ε, για μας από ό,τι τις χώρες που προσχώρησαν το 2004 ή το 2007 όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία και για την Κροατία. Και τώρα ε, για μας αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, όμως το μόνος τρόπος πρέπει να τα καταφέρουμε Ας ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, ε, τις πρωταξιακές διαδικασίες. Είμαστε ψηφία χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει καταντήσει ανέκδοτο πλέον. Είχαμε θετικές εκθέσεις που πλευρά της Επιτροπής η πρώτη του 2009. Και χάσαμε την ηθική μας πηξίδα περιμένοντας σε αυτή την αίθουσα αναμονής. Αποδείξαμε πως μια χώρα μπορεί να χάσει τη σειρά της αν αφαιρέσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική. Κινητοποιηθήκαμε, μεγαλώσαμε, βρήκαμε έναν τρόπο επικοινωνία με την αντιπολίτευση, όμως θα πρέπει να υπάρχει πάντα ευρωπαϊκή προοπτική. Και η επένδυση σε δημοκρατικά ευρωπαϊκά Βαλκάνια είναι πολύ μικρότερη αν αποφασίσουμε να την αγνοήσουμε. Γιατί τότε η επένδυση θα είναι τεράστια και σε οικονομικούς όρους και σε όρους ασφάλειας κτλ. Είναι ο μόνος τρόπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητάω συγγνώμη αν δεν απάντησα σε κάποια ερωτήματα, ίσως ένα-δύο να μην τα απάντησα. Την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ υπόσχομαι ότι θα φέρω περισσότερες ε, ε, πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αγαπητέ Υπουργέ, Νικόλα Δημήτρου, Μπορώ να πω εκ μέρου όλων των συναδέλφων στην Επιτροπή μα ότι σα ευχαριστούμε για την ενημέρωση για τι τελευταίε εξελίξει στη χώρα μα. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία και όχι μόνο ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, αλλά και ως ενεργό μέλος ε, της οικογένειας του ΕΛ και ως αντιπρόεδρος του κόμματο. Ε, θα ήθελα προσωπικά να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για αυτό το ζωτικό δημοψήφισμα τον επόμενο μήνα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ελαφρώς καθυστερήσει κατά 12 λεπτά, αλλά νομίζω ότι άξιζε να έχουμε μια πιο μακροσκυλή συζήτηση με τον Υπουργό. Τώρα θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ερχόμαστε στην έκθεση και θα ήθελα να δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Βάιγκλ, που είναι ο εισηγητής. Και Μήπως ε, μπορείτε να βγάλετε έξω τις φωτογραφίες εκτός της αιθούσης. Could I also ask the non... Να ζητήσω από τα μη μέλη της Επιτροπής να συνεχίσουν ε, τις συζητήσεις τους εκτός της αίθουσας, αν είναι δυνατόν. the Και εσείς, ε, κύριε, με την κόκκινη γραβάτα. Μήπως θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε τις συζητήσεις σας, μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε Βάγκλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, που καλέσατε τον Υπουργό είχαμε μια εξαιρετική εισαγωγή στη συζήτησή μας ε, σχετικά με την έκθεση. Θα είναι δύσκολο να προσθέσω κάτι στα επιχειρήματα που ακούστηκαν. Και από ό,τι καταλαβαίνω το πιο σημαντικό επιχείρημα και μάλιστα πετύχαμε μεγάλη ενότητα στην Επιτροπή μας είναι η ευρωπαϊκή προοπτική για τη Μακεδονία, ότι είναι σημαντική και είναι σημαντική για όλους μας. προκειμένου να έχουμε μια ασφαλή Ευρώπη. Προετοίμασα μια σύντομη ομιλία ως εισηγητής και θα την ε, υλοποιήσω χάρη της διαδικασίας, αν και δεν έχω κάτι ουσιαστικό να προσθέσω σε όσα υπόθηκαν την προηγούμενη μία ώρα. Να σας ε, πω λοιπόν ε, ότι η Μακεδονία όντως βρισκόταν στην αίθουσα αναμονής. για πάρα πολλά έτη. Και όταν τώρα συζητούμε το σχέδιο του ψηφίσματος το πράττουμε σε συνθήκες πολύ συγκεκριμένες για την υποψήφια χώρα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική ιστορική συγκυρία. Θέλω να αναφερθώ στη σημασία του δημοψηφίσματος της 30ης Σεπτεμβρίου. Με μεγάλη χαρά άκουσα τους συναδέλφους από το ΕΛΚ που ανακοίνωσαν ότι έχουν ε, διαφορετική θέση από το κύριο αντιπολιτευόμενο κόμμα της ε, Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι η αντιπολίτευση στη Μακεδονία θα ακολουθήσει αυτά που υποστηρίζουν ε, και τα αδελφά κόμματα το αδελφό κόμμα. Θέλω να επαναλάβω ότι και οι δύο διαπραγματευτές και από την Ελλάδα και τη Μακεδονία μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις ιστορικές παρεξηγήσεις και να προσφέρουν στις χώρες αλλά και σε εμά ένα πραγματικό μέλλον για την περιοχή και για όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Το ίδιο ισχύει και για την ε, διπλωματία και τις κυβερνήσεις ε, και την κυβέρνηση της Βουλγαρίας και της Μακεδονίας. Δημιουργήθηκε ένα νέο παράδειγμα για τις ε, μελλοντικέ σχέσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ευρώπη γενικότερα. Έχουν συνεισφέρει σε μια νέα φιλοσοφία διμερών σχέσεων. Η Μακεδονία θα πρέπει μετά το επιτυχές δημοψήφισμα, που ελπίζω να είναι επιτυχές, θα πρέπει να επανέλθει στο καθήκον της και να συνειδητοποιήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, το φιλόδοξο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, στο δικαστικό σύστημα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, στην προστασία των μειονοτήτων και άλλα ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το ρόλο του ειδικού εισαγγελέα και του ομπούτσμαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως υπόθηκε και στο παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια συνεχώς υποστήριζε την ε, ευρωπαϊκή και την ε, νατοκή προοπτική της ε, Μακεδονίας. Φυσικά αναμένω να συνεργαστώ με τους συναδέλφους που θα ήθελα να παρουσιάσουν τροπολογίες στην έκθεσή μου και θα έχω τη δυνατότητα να συνεργαστώ και με δημιουργικού και οδησυγητές από τα άλλα κόμματα. Ευχαριστούμε για τη σύντομη παρουσίαση τη εκθεσή σας. Τώρα έχουμε κάποιο χρόνο για την ε, πρώτη εξέταση. Ποιος ε, έχει ζητήσει το λόγο μέχρι τώρα, κανείς. Ήδη συζητούσαμε το θέμα της μακεδονία αλλά ίσως ο κύριος Πέτερ λέει να θέλει το λόγο ως ε, πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε σχέση με όσα ανέφερα στην προηγούμενη συζήτηση. Σαφώς έχει αλλάξει η κατάσταση, έχει βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά, αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Φυσικά είναι κάπως ε, σχετικά ήρεμες οι συνθήκες ε, διοργάνωσης του δημοψηφίσματος και χαίρομαι που μπορούμε να λειτουργήσουμε σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε ένα τέτοιο κλίμα. Βλέπω να υπάρχει ενότητα μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων και ελπίζω ότι αυτή η υποψήφια χώρα θα μπορέσει τελικά να βγει από την αίθουσα αναμονής. Κάτι που προκαλούσε και μεγάλη σύγχυση. Επίσης, ελπίζω ότι η κοινή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα λάβει χώρα στα Σκόπια σε ένα ευχαριστό κλίμα. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο, ο κύριος Κέλαμ. Ευχαριστώ. Ω σκιώδης εισηγητής για την έκθεση αυτή θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βάικολ για το κείμενό του. Νομίζω ότι μας διευκόλυνε πολύ η νέα Μακεδονική κυβέρνηση στο καθήκον μας και μπορούμε να συμπεράνουμε στην έκθεση αυτή ότι υποστηρίζουμε πλήρως τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση θα πρέπει να ξεκινήσουν του χρόνου. Φυσικά, πολλά θα πρέπει να γίνουν και όπως λέγεται και στην έκθεση της Κομισιόν, έχει επιτευχθεί πρόοδος σε πολλούς τομείς και στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, όμως πολλά απομένουν να γίνουν. Πιστεύω όμως ότι εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει οπισθοδρόμηση. Αυτό που είναι ανησυχητικό σήμερα πριν το δημοψήφισμα είναι ότι κάποια πολιτικά κόμματα όπως το ΒΜΡΟ έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στο δημοψήφισμα και στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως ε, την έκκληση του Έλμαρ Μπρόκ στο αδελφό μας κόμμα ότι θα πρέπει να λάβει μια θέση κάτι που αφορά τα συμφέροντα της χώρας συνολικά. Φυσικά θα κατατεθούν κάποιες τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι φέτος το έργο μας θα είναι πιο εύκολο και πιο παραγωγικό από ό,τι στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλεμ, ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βάικολ και εξ ονόματος της ομάδας μου για μια εξαιρετική έκθεση μας παρουσιάζει τα κύρια γεγονότα στην σημαντική περσίνη χρονιά. Η βελτίωση του πολιτικού κλίματος στη χώρα αλλά και η θέση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη Μακεδονία κατέληξαν σε μια πραγματική πρόοδο στη χώρα αυτή που περίμενε πάρα πολύ καιρό για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μακεδονία είναι πράγματι το πιο φωτεινό παράδειγμα πρόοδου όχι μόνο μεταξύ των ε, χωρών ε, που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ένωση, αλλά είναι και ένα σπάνιο παράδειγμα επιτυχούς ε, εφαρμογής της στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε που η κυβέρνηση έχει βελτιώσει και τις σχέσεις της ε, με τους γείτονες, αλλά υπάρχουν και σημαντικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Το πολιτικό κλίμα στη χώρα κατέστησε δυνατό να βελτιωθούν οι σχέσεις ε, μεταξύ των διάφορων ε, εθνοτήτων και να υπάρξει και καλύτερος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Φυσικά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη σε ό,τι αφορά την μεταρρυθμίση του δικαστικού συστήματος, τη μεταρρυθμίση των μυστικών υπηρεσιών, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης υπάρχει και πρόβλημα με την παραοικονομία. Και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα πρόοδου. Όμως το πιο σημαντικό είναι το δημοψήφισμα και η σχετική εκστρατεία. Η συμφωνία που επιτεύχθη με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για το μέλλον της χώρας αλλά και ολόκληρης της περιοχής ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Η κυβέρνηση αυτή μας έχει δείξει ότι έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει τα πιο δύσκολα προβλήματα. Θέλουμε να προσφέρουμε την υποστήριξή μας στη Μακεδονία και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δούμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων και να την καλωσορίσουμε στην επόμενη εκθεσή μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Πίτσουλα. Από το ΙΣΙΑΡ δεν θέλει κανείς το λόγο, ούτε από το ΑΛΔΕ ή από τους Πρασίνους. Παρακαλώ, κύριος Μεζέρτης, από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρέντα, για το σχόλιο. Όταν ανέλαβα τη θέση του σκιώδου συζητητή, δεν μου είχε περάσει καλά από το μυαλό ότι ολόκληρη την πολιτική μου, σε ολόκληρη την πολιτική μου καριέρα θα φτάναμε σε ένα σημείο που τελευταία πρόταση της έκθεσης δεν θα ήταν απλώς ε, μία αόριστη ελπίδα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση χάρη στη διπλωματία και χάρη φυσικά στον εισηγητή. Ε, το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό και τον ευχαριστώ. Θα στείλουμε κάποιες ε, τροπολογίες που θα είναι όμως τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν τα συνήθη θέματα τι μεταρρυθμίσει που έχουν να αντιμετωπίσουν όλε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, κατά πολέμηση τη διαφθορά, δικαστικό σύστημα κτλ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να τονίσω ότι ένα από τα κύρια σημεία για αυτό το δημοψήφισμα θα είναι παραδείγματο χάρη, μια δοκιμή για την ελευθερία και τον πλουραλισμό των την πολυφωνία των μέσων μαζική ενημέρωση. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να χειριστεί κανείς ε, τα ΜΜΕ με έναν επικοδομητικό και νόμιμο τρόπο σε μια ε, πιθανά τεταμένη ε, εκστρατεία. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και σε σχέση με το αν θα έχει επιτυχία το δημοψήφισμα. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή να ζητήσει και από την πολιτική του ομάδα να στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία αντιπροσωπεία για το δημοψήφισμα. Θα πρέπει να ε, στείλουμε μία πλήρη αντιπροσωπεία παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρατηρήσει το δημοψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Ένταξε. Ρώτησα και τη γραμματεία αν έχει ληφθεί απόφαση για την αποστολή αντιπροσωπείας από το Κοινοβουλίο. Θα το ελέγξω, συνάδελφε. Είναι σημαντικό. Ωραία. Η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή τον κύριο Βάγγελ, για, την, ε, για το καλό κείμενο που έχει ολοκληρώσει και φυσικά πάνω σε αυτό το κείμενο όπως κάθε φορά θα κάνω και εγώ κύριε Βάγγελ, τις ε, δικές μου βελτιώσεις όπως κάθε χρόνο. Ε, γνωρίζουμε όλοι κάτω από ποιε συνθήκε και από ποιε μεθοδεύσει φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση στη Φύρο. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο χρόνο και κάτω από δύσκολε συνθήκε έχει κάνει θετικά βήματα σε αρκετού τομεί. Υπενθυμίζω όμω ότι για τους λόγου που προανέφερα γινόταν προσπάθεια ωρεοποίηση τόσο καιρό και στρογγυλοποίηση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα, δίνοντα έτσι περιθώριο αλλά και χρόνο στο προηγούμενο καθεστώ να δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία απήχε πάρα πολύ από τα κριτήρια αλλά και από όλες τις προϋποθέσεις για μια ομαλή ενταξιακή πορεία. Υπενθυμίζω ότι το συστημικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Γκουρεύσκη οξύνθηκε σημαντικά με την πολιτική κρίση των τελευταίων χρόνων και ενισχύθηκε από αυτή την πολιτική τακτική για την οποία είναι υπεύθυνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρεώνοντας σε τρίτες χώρες τα προβλήματα που υπήρχαν στη χώρα και όχι στους ίδιους τους πολιτικούς της χώρας. Όμως, ε, κύριε Βάγκλη, στάση αυτή έχει και ένα θετικό, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για μένα και το οποίο στα τέσσερα χρόνια που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πρώτη φορά που το, το παρατηρώ. Ε, δεν χρησιμοποιήσατε από πουθενά στο κείμενό σας τη λέξη Μακεδονία, για το οποίο αρκετές φορές είχα κάνει τροπολογίες, τις οποίες δεν είχατε αποδεχτεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου εξηγήσετε για αυτή, γιατί αυτή η διαφοροποίηση από τα προηγούμενα κείμενα στα τώρα. Έχει και θετικό γεγονός, και ένα ακόμη, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Τώρα η προσοχή της χώρας δεν θα αποσπάται από τις δικαιολογίε που έβαζε μέχρι τώρα στην αποτυχία της να δεσμευτεί σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, τις οποίες αναφέραμε και δεν χρειάζεται να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Τώρα για τη χώρα είναι η στιγμή που θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για μεταρρυθμίσεις και να τις ολοκληρώσει για να ενταχθεί αν θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντα, θα ήθελα να σημειώσω και να πω το τελευταίο. Διαφωνώ με όσους θεωρούν ότι η γρήγορη έναρξη των διαπραγματεύσεων θα δώσει παραπέρα κίνητρα για εκδημοκρατισμό και θα ενισχύσει τον έλεγχο, τη λογοδοσία και τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς τις μεταρρυθμίσεις αν οι ίδιοι δεν θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Πρώτα πρέπει να το θέλουν αυτοί και εμείς θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Όχι εμείς να το θέλουμε και εκείνοι να προσπαθούν ή να μην θέλουν να το κάνουν. Αυτό και ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστούμε την κυρία Σακοράφα. Δύο ακόμα ομιλητέ. Ο κύριος πρώτος. Thank you, Chair. I will speak in Greek. Uh, η πρόσφατη συμφωνία των κυβερνήσεων Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν, ε, δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των λαών των δύο χωρών και των υπολείπων λαών της περιοχής. Προωθείται με την ξεκάθαρη και απροκάλυπτη παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τις ε, δύο κυβερνήσεις με σκοπό την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα βήμα ολοκλήρωσης των ε, Βαλκανίων, μιας περιοχής κλειδί για τους ανταγωνισμούς που αναπτύσσονται και είναι πολύ σφοδροί ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις και τη Ρωσία και την Κίνα. Η κίνδυνη είναι μεγάλη. Η παρουσία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή είναι εχθρική για την ασφάλεια των λαών και συνδέεται με αφισβητήσει συνόρων, παραβιάσει κυριαρχικών δικαιωμάτων, ανακίνηση υπαρκτών και ανύπαρκτων μειωνοτικών ζητημάτων, ενίσχυση των στρατιωτικών βάσεων. Χαρακτηριστικό είναι επίση το στοιχείο τη ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων, που ε, ένα από αυτά είναι η προώθηση των αντεργατικών, των σκληρών αντιλαϊκών μέτρων στο όνομα των μεταρρυθμίσεων των λεγόμενων, με ειδικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου και αυτής της απαράδεκτης έκθεσης που ε, του ψηφίσματος που προωθείται εδώ. Ε, ακόμα και στο ζήτημα της ονομασίας της ε, ε, χώρας, η συμφωνία παραπέμπει στο αβέβαιο μέλλον και διαιωνίζει σπέρματα αλυτρωτισμών για τη γλώσσα, για την εθνικότητα που υποδαβλίζονται και αξιοποιούνται από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όπω έχει δείξει τόσο η πείρα με τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία, όσο και οι προεθούμενες αλλαγέ συνόρων μεταξύ Σερβία και του προτεκτοράτου του Κωσόβου. Η συμφωνία λοιπόν δεν εξασφαλίζει την ειρήνη, τη συνεργασία και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Αντίθετα, αποτελεί κίνδυνο για του λαού ε, τόσο των δύο χωρών όσο και της ευρύτερης περιοχής και γι' αυτό χρειάζεται σήμερα επαγρύπνηση και πάλι να μπουν ε, και πάλι για να μπουν εμπόδια σε όλα αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα, εξ ονόματος ε, του κυρίου Κούκαν, παίρνω το λόγο γιατί δεν βρίσκεται εδώ σήμερα. Ήθελε όμως ε, να μεταφέρει ένα μήνυμα που λέει ότι η Μακεδονία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ε, και έχει επανέλθει στον ευρωατλαντικό δρόμο. Αναγνωρίζουμε την προσήλωση της νέας κυβέρνησης σε αυτή τη διαδικασία, καθώς ε, και τα συμπεράσματα Συμβουλού και Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανοίγουν το δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων το 2019. Τονίζουμε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να σημειώνουν πρόοδο και να δημιουργήσουμε όθηση για την επιτυχή έναρξη των διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο του 2019. Αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε τις προσπάθειες ε, της κυβέρνησης για την προώθηση των αγαστών σχέσεων με τις γειτονικέ χώρες, ιδίως με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Θετικές εξελίξεις, ελπίζω, λέει ο κ. Κούκαν, οι Μακεδόνες να υποστηρίξουν την συμφωνία με την Ελλάδα στο επερχόμενο δημοψήφισμα θα είναι κρίσιμα σημασία για τον μελλοντικό προσανατολισμό της χώρας. Το πολιτικό κλίμα στη χώρα έχει αλλάξει Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευμερία, της σταθερότητα και την ανταξιακή διαδικασία. Πρέπει να ενισχύσει τη δημοκρατική διαδικασία και το κράτος δικαίου. Είναι σημαντικό οι συνεχιζόμενες αυτές θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις να γίνουν με ένα ανοιχτό και δημοκρατικό τρόπο, με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα για το κράτος δικαίου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθούν οι κρίσιμες ε, και οι επίγουσες ε, προτεραιότητες σε φορά τις μεταρρυθμίσεις. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ανακτήσει το ρόλο του στην ε, δημοκρατική εποπτεία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται ότι πάντα είναι διατεθειμένο να στηρίξει ε, και να παράσχει κάθε συνδρομή στη Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο του διαλόγου Ζαν Μονέ και στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών για την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Τέλος. Είναι θετική η έκθεση που δείχνει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαδικασίες μεταρρύθμισης και τη διαδικασία της ε, ένταξης αυτής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, Κρίστιαν. Άλλος, κανείς, όχι. Να δώσουμε το λόγο στον Γενικό Διευθυντή για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, εξότιμα μέλη, ε, αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Βάγκλ για το σχέδιο ψηφίσματος και για όλο το έργο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και με τους βουλευτές Φλέκενσταν και Κούκαν για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας και για τη διεξαγωγή του διαλόγου Ζαν Μονέ. Είναι αυτά παραδείγματα για το πώς το Κοινοβούλιο προάγει τις δημοκρατικές διαδικασίες σε όλες τις χώρες. Είπατε πολύ σωστά ε, ότι η χώρα αυτή έχει υπερβεί πλέον, έχει ξεπεράσει την πολιτική κρίση και έχει επανέλθει στον δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και η κυβέρνηση, ο κύριος ε, Υπουργός μάλλον, η κυβέρνηση έχει σημειώσει σημαντικά βήματα για την βελτίωση των σχέσεων με γειτονικέ χώρες ε, και με τη διμερή συμφωνία με την Βουλγαρία και με την συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτή η ιστορική συμφωνία είναι ένα παράδειγμα και υπόδειγμα για την περιφέρεια και για την Ευρώπη εν γέννη. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες με όλα τα μέσα. Είναι μια μοναδική ευκαιρία το επερχόμενο δημοψήφισμα για τους πολίτες να αποφασίσουν το μέλλον της χώρας τους. Ο δρόμος είναι σαφής. Είναι ο δρόμος προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλες οι πολιτικές ε, ε, δυνάμεις πρέπει να αναλάβουν ε, τις ευθύνες τους, να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες και προσδοκίες των πολιτών και να ανταποκριθούν στο όραμα της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης. Και στην περασμένη έκθεση είπαμε ότι η μεταβατική προσωρινή συμφωνία έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και έχουν υλοποιηθεί οι ε, βασικές μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό και συστήνουμε εμεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων και τον Ιούνιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και άνοιξε το δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο του 2019 πρέπει να διατηρήσουμε την ε, σημερινή όθηση που υπάρχει και δυναμική για την ε, υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, ιδίως σε τομείς όπως ο δικαστικός ε, τομέας, οι μυστικές υπηρεσίες και η δημόσια διοίκηση. Τέλος, ε, να επισημάνω ότι με προσήλωση εμείς ε, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες μεταρρύθμισης αυτής της χώρας και στηρίζουμε τις ανταξιακές της προσπάθειες. Ο Επίτροπος Χάν επισήμως έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου στα Σκόπια τον Ιούλιο με ιδιαίτερη έμφαση στα κεφάλαια που άπτονται του κράτους δικαίου θα ε, πάει και πάλι στα Σκόπια σε μερικέ εβδομάδε και ο Κρίσταν Ντάνιελ, Γενικό Διευθυντή, βρίσκεται σήμερα στα Σκόπια. Αυτέ είναι μερικέ μόνο ενδείξει για την ε, σημαντική προσήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές προοπτικές αυτής της Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στον εισηγητή για τα καταληκτικά του σχόλια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να προσθέσω ότι πράγματι τα περασμένα χρόνια που αντιμετωπίζαμε μια πολιτική κρίση στη Μακεδονία, παρόλα αυτά υπήρχε εξαιρετική συνεργασία και κατανόηση μεταξύ του Κοινοβουλίου μας και της Επιτροπής. Και πρέπει να αναγνωρίσω και την ε, προσωρινή δέσμευση και εφευρετικότητα σε ό,τι αφορά την επίλυση δύσκολων προβλημάτων. Και αυτό μας οδήγησε στην Συμφωνία Πρέτζινα. Ο Επίτροπος Χάν, λοιπόν, ε, συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, στα θετικά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα και το αναγνωρίζουμε. Άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον ε, όλες τις παρατηρήσεις σας, τις σημειώνω και ε, φυσικά και θέλω να συνεχίσουμε το κοινό μας έργο για την διαμόρφωση αυτής της έκθεσης και αποκοινούμε τους κοιόδες. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Ιβο Βάγκλ και τους συναδέλφους για τα σχόλια. Κλείνει η πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 6 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί. Και μετά θα περάσουμε στη δεύτερη εξέταση στις 27 Σεπτεμβρίου εδώ στην ΑΦΕΤ. Περνάμε τώρα στο σημείο 6. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 18 για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Να δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον μοναδικό Κρίστιαν Πρέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Χαίρομαι που μπορώ να παρουσιάσω σήμερα την τέταρτη έκθεση που για τη η Ερτσεγοβίνη. Πόσο μάλλον που σήμερα το απόγευμα θα επισκεφτώ το Σεράγεβο μαζί με κάποιους συναδέλφους στα πλαίσια της αποστολής του ΕΛΚ που οργανώθηκε από τον Αντρέν Κόβατσεκ. Επίσης, έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την πρώτη το πρώτο σχέδιο στα μέλη της Βασίλισσας Ενωμένης, στα μέλη του Συμβουλίου και στα μέλη των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Καθώς την επόμενη μέρα των συζητήσεών μας θα έχουμε τη δυνατότητα να τους αναφέρουμε απευθείας το τι συμπεριλαμβάνει η έκθεση αυτή. Θέλουμε να περάσουμε διάφορα μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό μέλλον τη Βοσνία Ερσεγοβίνη και θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη χώρα αυτή. Έτσι λοιπόν, ε, όταν είχαμε την επίσκεψη του Πρόεδρου Γιούγκη στο Σεράγεβο ε, το Φεβρουάριο και απαντήθηκε το κατάλληλο ερωτηματολόγιο, είναι κάτι που το χαιρετίζουμε. Χρειάστηκαν 15 μήνε οι αρχέ και ελπίζω ότι πρόσθετε απαντήσει απαντήσεις να μπορούν να δοθούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, μας ανησυχεί η μεγάλη καθυστέρηση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων λόγω των πολιτικών διαφορών που εμφανίστηκαν κατά την προεκλογική εκστρατεία που ξεκίνησε πάρα πολύ νωρί ακόμη και για τα στάνταρ τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που πάντοτε ξεκινούσε την εκλογική διαδικασία αρκετά νωρί. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι παρά την απουσία συμφωνίας ε, για τον εκλογικό νόμο θα πρέπει οι εκλογές του Οκτωβρίου να υλοποιηθούν σε καλές συνθήκες και θα πρέπει το αποτέλεσμα ε, να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως. Ε, περιμένουμε το ελάχιστο από μια υποψήφια χώρα, δηλαδή να ελοπίσει τις εκλογές και να θέσει σε εφαρμογή το αποτέλεσμα. Να ελοπίσει το αποτέλεσμα είναι μια πρώτη απέτηση για κάθε χώρα που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο μήνυμα είναι ότι μετά τις εκλογές οι αρχές θα πρέπει να συσταθούν εντάχει και όλοι οι πολιτικοί φορείς θα πρέπει να ε, αγωνιστούν ε, για την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων έχοντας ε, ως στόχο την ένταξη στην Ένωση. Μεταρρυθμίσεις κοινωνικές και οικονομικές αλλά όχι μόνο γιατί η χώρα χρειάζεται πάρα πολλές αλλαγές. Στο σχέδιο έκθεσης υπάρχει ένας μακρύς ε, κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα κατά πολέμηση της διαφθοράς, ενίσχυση του κράτους δικαίου και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης, μεταρρύθμιση της δημοσίας διοίκησης φέτος ε, επέμενα ιδιαίτερα στο θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναφέρω εδώ την αναγκαιότητα να αναλυφθεί δράση ως προς τη μη εισαγωγή διακρίσεων. Επίσης υπάρχει αναγκαιότητα να σταματήσουν διακρίσεις κατά των πολιτών που έχουν διαπιστωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβουργού καθώς ε, και κάθε άλλη μορφή διάκρισης. Επίσης, ε, αναφέρω την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ε, πρόσφατα είχαμε το προηγούμενο ε, Σαββατοκύριακο ε, επίθεση κατά του δημοσιογράφου Κοβάσεβιτς και το 61% συγγνώμη, 61 δημοσιογράφοι, σύμφωνα με την Ένωση Δημοσιογράφων, ε, δέχτηκαν επίθεση ε, το 2017 και 41 ε, το 2018. Είναι ανησυχητικό. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα και θα πρέπει οι πολιτικοί να εργαστούν για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον προκειμένου να μπορούν οι δημοσιογράφοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτά είναι τα κύρια μηνύματα που θα συγκρατούσα εγώ και φυσικά θα ήθελα να ακούσω και τους συναδέλφους. Είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία μας θα είναι πολύ καλή όπως και τα προηγούμενα έτη για την εκπόνηση της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Christian, for your Ευχαριστώ. Κριστιαν για την παρουσίαση. Να δώσω το λόγο, το λόγο πρώτα στον κύριο Πίτσουλα, πρόεδρο της ε, αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πρέντα για την εξαιρετική έκθεση η οποία συνοψίζει τις εξελίξεις στην Βοσνία και Εργοβίνη τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και ο επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας του ΕΕΛ και καλωσορίζω το γεγονός ότι, ότι στο επίκεντρο είναι το ανεπίλητο θέμα ότι η κοινή κοινοβουλευτική ε, συνέλευση δεν έχει ε, συνέλθει τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε θέματα που φορούν ε, το περιβάλλον, το δίκαιο. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδο το τελευταίο χρόνο. Υπάρχει τελμάτωση και ενώπιση των εκλογών του Οκτωβρίου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Βλέπουμε ότι η εκστρατεία του Τούρκου Προέδρου επικεντρώνονται στη γενοκτονία, αλλά εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία για την ε, ευθυγράμμιση του εκλογικού νόμου με την απόφαση του δικαστηρίου, όλα αυτά είναι θέματα υποσυζήτηση. Κάνουμε λόγο για την ε, εκπροσώπηση των πολιτών από άλλες εθνοτικές ε, κοινότητες. Σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να έχουμε μια ρήτρα η οποία θα αναφέρει την βασική αιτία όλων των προβλημάτων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το γεγονός ότι η συμφωνία του Ντέιτον δεν λειτουργεί. Αν την τροποποιήσουμε, ίσως να έχουμε ε, σωστή λειτουργία με βάση το κράτος δικαίου, την αρχή της επικουρικότητας και να εγγυηθούμε την ε, επαρκή εκπροσώπηση των κοινωτήτων και των πολιτών. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και ανυπομονώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Tonino. Ευχαριστώ τον Νίνο. Τώρα περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Ζούιτσα έχει στήσει το λόγο. Κυρία Ζόφκο. Από το S&D. Να σημειώσουμε τα ονόματα. Ζόφκο. Από το ECR. Δεν θέλω να με κατηγορήσετε και πάλι ότι δεν σημειώνω αυτά τα ονόματα, γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον κατάλογο των ομιλητών. Μπέλντα, από το ECR, να μην κάνουμε λάθος. Κύριο Σεράντος, στη συνέχεια, από τους πρασίνους όχι. Γκουε. Ο κύριος Κόλιτσεκ δεν είναι εδώ, FDD. Καστάδο δεν είναι εδώ. Δεν έχουμε άλλους. Ζήτσα Ζόφκο, Παπαδάκης, Μπέλτα Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Παπαδάκη. Συγητή είναι ισορροπημένο και αγγίζει τα πιο σημαντικά θέματα που καλούμαστε να εξετάσουμε αναφορικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Βοσνία Ζεβοβίνη. Θεωρώ ωστόσο πως σε ορισμένα σημεία οι σχετικές διατυπώσεις χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Θα καταθέσουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες. Καταρχήν πρέπει να αναδείξουμε και να τονίσουμε ακόμη περισσότερο ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας θα αλλάξει τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Θα επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί πολιτεύονται, και θα δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον σε όλους τους πολίτες της χώρας, ανεξάρτητα από την εθνική προέλευση ή τη θρησκεία τους. Πρέπει να διασφαλιστεί πλήρης και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ατζέντα μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε από τις αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης προς όφελος των πολιτών της και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρει και ο εισηγητής, εκφράζω και εγώ με τη σειρά μου την ικανοποίηση για την οριστικοποίηση των απαντήσεων της χώρας στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, αλλά παράλληλα πρέπει να ανταποκριθεί έγκαιρα και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πρέπει να τονιστεί η ανάγκη οθέτησης ενός στρατηγικού προγράμματος για τη σταδιακή ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό γεχτημένο, μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό και συντονισμό. Σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει για την εμπλοκή του στην ενταξιακή διαδικασία. Δεν παρατηρηθήκε πρόοδο στην ελευθερία έκφραση και στην οικοδόμηση ανεξάρτητων μέσων ενημέρωση. Η εναρμόνιση τη χώρα με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη βελτιωθεί. Η ικανότητα διαχείρισης της μετανάστευσης, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση ευάλωτων ομάδων, πρέπει να ενισχυθεί. Η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων είναι ζήτημα κέρια σημασίας, καθώς δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και στους Ρωμά σε σχέση με τις κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσέγγισης με μεγαλύτερη έμφαση στο κοινωνικό σκέλος. Όλες οι εμπλεγόμενες πλευρές θα πρέπει να σκεφτούν το κοινό όφελος των πολιτών και οι γειτονικέ χώρες πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό. Βεβαίως όμως πολύ σωστά υπογραμμίζει και ο εισηγητής, οι δυσκολίες παραμένουν και χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά και έμπραχτη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Αυτά προς το παρόν από τη δική μας πλευρά. Ευχαριστώ τον εισηγητή και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία όπως άλλωστε είχαμε και τη χρονιά που μας πέρασε. Thank you. We now come Ευχαριστώ στον κύριο Μπέλντερ και όδη από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε Πρέντα, σας ευχαριστώ θερμά για την ξεκάθαρη αυτή έκθεση για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. ω ε, και πρώην δημοσιογράφο. Ε, θεωρώ εξαιρετικά σημαντική αυτή την παράγραφο ε, για την ελευθερία στον τύπο. Κάνατε και μία ιδιαίτερη μνήμα στην στην δειλή αυτή, η θρασίδηλη επίθεση προς τον δημοσιογράφο Κοβάτσαβιτς και πολύ σωστά αναφέρατε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ε, σχέση ε, και ε, με τη μεταφορά ειδήσεων από το Σαράγεβο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διασφαλίσουμε την ελευθερία του τύπου. Κάτι ακόμα που θέλω να επισημάνω, γιατί το θεωρώ σημαντικό, είδα ότι στην έκθεση δεν γίνεται λόγος για την επιρροή τρίτων εξωτερικών δυνάμεων στη Βοσνία, το οποίο είναι σημαντικό θέμα, που προσελκύει το ενδιαφέρον. Φυσικά εδώ έχουμε να κάνουμε με τη Ρωσία, ε, με τη Ρεπούμπλικα Σρεύσκα, αλλά και με άλλες ε, οντότητες, και η Τουρκία και οι χώρες ε, του κόλπου έχουν επιρροή και εσωτερικά και εξωτερικά και στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημά μου είναι, ποια είναι η δική σας θέση προς τους ε, εξωτερικούς αυτούς παράγοντες. Ο Κόναντ Άντενάουερ ε, αναφερόταν σε αυτό στο παρελθόν και εγώ το είχα επισημάνει ότι υπάρχει αυτή ε, η παράληψη. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί κάτι εδώ. Πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και περνάμε στον κύριο Ράντος για το Άλντε. Θέλω να ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Πρέντα για την ολοκληρωμένη έκθεση, για την προσφορά του θα αναφερθώ στα πιο κέρια ζητήματα και είναι αποτυχία επίτευξη συμφωνία για τον εκλογικό νόμο για τη Βουλή των Λαών, όχι μόνο στην Ομοσπονδία αλλά και στην Σερβική Δημοκρατία. Η κατάσταση είναι πολύ χειροτερή στην ε, Σερβική Δημοκρατία. Η ψηφία εξυπηρετούν ε, τα συμφέροντα της πλειοψηφίας από, τη, από την μειοψηφία. Η Βουλή των Λαών είναι ένας θεσμός ο οποίος προβλέφθηκε από τη συμφωνία του Ντέιτον και προστατεύει τα δικαιώματα και των τριών εκλογικών περιφερειών, αλλά δεν εκπροσωπούνται τα συμφέροντα των κοινωνικών των μειονοτήτων και αυτό δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και παρεμποδίζει την πρόοδο σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης, τα δικαιώματα των μειωτητών και την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι ένα πρόβλημα και θεωρώ ότι θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο στην έκθεση. Οι τροπολογίες μας θα κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Ράντος. Δεν έχουμε άλλα αιτήματα από τις άλλες παρατάξεις. Συγχαρητήρια στον κύριο Πρέντε για αυτή την έκθεση. Είναι αντικειμενική και ολοκληρωμένη, όμως οι εκλογές, η προσεχή του Οκτωβρίου θα παρεμποδίσουν τη μελλοντική πρόοδο. Κάνω λόγο για την εξαρτή συγκεκριμένα. Ο κύριος Πρέντε κατονόμασε όλες τις, όλες τις τομείς στις οποίες δεν έχει σημειωθεί πρόοδος και αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον κύριο Πίτσουλα απέτυχε να περάσει το καταστατικό αυτό απεικονίζει την κατάσταση στη Βοσνία Ζεργοβίνη και κατά πόσο καταφέραμε να καταφέρουμε κάτι. Δεν πετύχαμε συμφωνία και είναι κρίμα. Κάνουμε λόγο και για τις εξωτερικές επιρροές. Ξέρουμε ποιοι επηρεάζουν την κατάσταση. Είναι παρούσα εξωτερική επιρροή, αλλά όλα εξαρτώνται από το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση ή εντός της χώρας. Δεν είναι ληστικό να ε, αναμένουμε μια υπεύθυνη στάση εν ώψη των εκλογών, θεωρώ ότι αποτυχία να εφαρμοστεί η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την υπόθεση Λιούμπιτς. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα εφαρμοστούν τα αποτελέσματα μετά τις εκλογές, θεωρώ ότι θα ε, δημιουργήσει πιο πολλά εμπόδια. Η Βοσνία Γοβίνη δεν έχει σημειώσει πρόοδο, έχει οπισθοχωρήσει και όσοι λένε ότι η συμφωνία του Ντέιτον πρέπει να πάνε να προσδιοριστεί. να έχουμε διατηρήσει ό,τι θέλουμε τελευταία χρόνια. Θέλουμε το κράτο Βοσνία Ζεγοβίνη και το, η αρχή τη επικουρικότητα θα πρέπει να παραμείνει βασική αρχή για τη λειτουργία του κράτου. Θα ταξιδέψω κι εγώ στο Σεράγεβο σήμερα ως μέρος της αποστολής εκ μέρους του ΕΛΚ και ελπίζω να συναντήσω τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη Βοσνία Ζεγοβίνη και να μπορέσω να λάβω απαντήσεις ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε κάποιες ε, τροπολογίες για να βελτιώσουμε την έκθεση του κυρίου Πρέντα. Ευχαριστώ. Κυρία Ζάφκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά για να μην χαθώ στη μετάφραση. Να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, τον κύριο Πρέντα, για αυτή την έκθεση. Εξαιρετική. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία τελευταία 23 χρόνια μετά τον πόλεμο η Βοσνία Ζεγοβίνη δεν έχει προχωρήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το απεικονίζει αυτό στα ψηφίσματα από το 2014. Το Διεθνής Ομάδας Κρίσης και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε μια αναλυτική έκθεση του 2017 ε, και με ψηφίσμα τον Ιανουάριο τα καταδεικνύει όλα αυτά. Θα πρέπει να στηρίξουμε πλήρως την έκθεση όπως και πέρσι. Έχει κάνει κάποιες στάσεις η Επιτροπή, όμως θα πρέπει να κάνει περισσότερα. Το να σιωπούμε σε μη αποτελεσματικέ πολιτικές δεν βοηθάμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βοσνία Ζεγοβίνη χρειάζεται περισσότερες ευρωπαϊκές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όπως είναι τα δικαιώματα των ε, κοινοτήτων, ε, ομοσπονδικός χαρακτήρας και η δημοκρατική εκπροσώπηση. Η Επιτροπή δεν πρέπει να λαμβάνει ε, το μέρος ε, μίας από τις ε, τρεις ανταγωνιστικές περιφέρειες. Μια τέτοια πολιτική θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αξιόπιστη. Μπορούμε να προτείνουμε στους ηγέτες των τριών κοινοτήτων να βρουν λύσεις μεταξύ τους. Αν η Βοσνία Ζεγοβίνη θέλει να επιβιώσει και κάποια μέρα να ε, δρέψει τα ωφέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χακλάιτνα, άλλη μια φορά από την ε, Digineer. Ευχαριστώ και πάλι, αγαπητά μέλη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για το σχέδιο έκθεσης. Θεωρούμε ισορροπημένο το κείμενο και σύμφωνο με τα πορίσματα της Επιτροπής από την έκθεση του 2018. Αυτή η έκθεση ήταν μια διάμεση έκθεση για τη Βοσνία Ερτζεγοβίνη για να παρέχουμε ενημέρωση για την κατάσταση στη χώρα, εστιάζοντας κυρίως στο κράτος δικαίου, τη δημόσια διοίκηση και τη μεταρρύθμιση και τις οικονομικές εξελίξεις. Πλήρης ανάλυση σε σχέση με τα κριτήρια προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνοδεύει αναλυτικές εκθέσεις και είναι μια συνεχόμενη διαδικασία η επίθεση στους δημοσιογράφους, του δημοσιογράφο καταδικάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την αντιπροσωπεία της εκεί. Είναι σημαντικό η Βοσνία Τσεγοβίνη να συνεχίσει να είναι αποδοτική στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, όσον αφορά τα κρατοδικεία, τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα, την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλα μπορούν να γίνουν πριν από τις εκλογές ε, της 7ης Οκτωβρίου, ε, όπως ε, ε, σημεία συνεργασίας με την ε, Europol. Συνεργασία και συντονισμός στη χώρα θα πρέπει να επίσης να ενισχυθεί να χρησιμοποιηθεί ο μηχανός PIH, για το συντονισμό όσον αφορά τη μετανάστευση. Τον Αύγουστο λήφθησαν διάφορες αποφάσεις από την Επιτροπή να παρέχουμε περαιτέρω ενίσχυση ε, στην Βοσνία Γοβίνη για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Διατέθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ, ε, τα οποία συμπληρώνουν τα 1,5 εκατομμύρια ε, που ε, προσφέρθηκαν τον Ιούνιο για την διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης. Όσον αφορά την εκλογική μεταρρύθμιση, είμαστε ξεκάθαροι ότι ε, η απόφαση εναπόκειται στην Βουλή των Λαών. Και η Επιτροπή Χάν και η κυρία Μογγενή ήταν ξεκάθαρη στις δηλώσεις της. Οι προσπάθειες διευκόλυνσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα έχουν παράσχει ένα πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει ε, σε μια λύση για τις εκλογές. Να τονίσω ότι η Επιτροπή είναι δεσμευμένη όσον αφορά τη Βοσνία Ζεργοβίνη, θα συνεργάζεται με τη χώρα και με διεθνείς οικονομικούς φορείς για την εφαρμογή της, ε, του θεματολογίου για την ε, ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ξαναδώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους καταρχήν που είναι παρόντες. Δεν είναι εύκολο μετά τις διακοπές. Επίσης, ε, κυρίως σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια σημεία. Αυτά που αναφέρω κύριο Σπιτσούλα, καταρχήν, την πρόσφατη απόφαση του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης της Μπανιαλούκα να ακυρώσει την έκθεση της γενοκτονίας της Εμπρένιτσα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για την προεκλογική όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια επίσημη πράξη αυτής της οντότητας, αυτού του φορέα. Είναι λοιπόν πραγματικά πολύ σοβαρό να υπάρχει επαναχώρηση στην έκθεση αυτή. Νομίζω έχουν περάσει ήδη 14 χρόνια. Το 2004 νομίζω αναγνώρισαν τη γενοκτονία. Η επαναχώρηση αυτή λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σημεία που αναφέρθηκαν από το συνάδελφο Παπαδάκη και συγκεκριμένα σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου και τα λοιπά σημεία που έθεσε. Όλα αυτά τα ζητήματα ήδη είναι υπό εκπόνηση ως τροπολογία στην έκθεσή μου, γιατί αυτά αποτελούν τμήμα της έκθεσης. Όμως, ε, ξέρετε, εδώ έχουμε κάποιους ε, κανόνες που πρέπει να συμβεστούμε σε σχέση με την έκθεση του κειμένου. Δεν ε, μπορούμε να έχουμε παρά ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων. Έτσι, λοιπόν, αυτά που ήθελα να βάλω στην έκθεση έπρεπε δυστυχώς να τα περιορίσω. Πάντοτε, έτσι είναι. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η εμπειρία από μια σκοπιά πνευματική, αλλά τέλος πάντων πρέπει να περικόψει κανείς διάφορα και στη συνέχεια να τα επανεισάγει ως τροποποίησης, ως τροπολογίες. Έτσι. Πρέπει να δουλεύουμε, τι να κάνουμε, πρέπει να σεβόμαστε όλους αυτούς τους νόμους, γιατί όλοι οι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται με την ίδια επιμέλεια. Τώρα, για τα θέματα που αναφέρθηκαν από τον συνάδελφο Μπέλτερ. Συμφωνούμε για τα όσα υπόθηκαν για την ελευθεροτυπία. Αυτά δεν συνδέονται μόνο με, τις πρόσφατες, με τα πρόσφατα γεγονότα. Δυστυχώς σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ο τύπος ε, υποφέρει. Ε, λόγω διάφορων ε, βιοπραγιών κατά των δημοσιογράφων. Επίσης, ε, πολιτικοί χρησιμοποιούν ε, τον τύπο ως ένα πολιτικό εργαλείο, όχι ως ένα εργαλείο για τους πολίτες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των ε, εξωτερικών πρωταγωνιστών. Και αυτό ήταν μέρος της εκθεσής μου και έπρεπε να το διαγράψω. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένως σε αυτό το θέμα και βέβαια όλοι όσοι αναφέρθηκαν, ε, Ρωσία, Τουρκία, τα κράτη του κόλπου, έχουν ε, μεγάλη παρουσία στη Βασιλεία Ερζεγοβίνη. Επίσης, ε, εδώ θα έκανα και μία επισήμανση, γιατί υπάρχουν ε, και διαφορετικές στάσεις. Οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, παραδείγματος χάρη, αναγνωρίζουν την επιρροή που ασκούν στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ρωτήσετε τον Πούτιν ή τον Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών, ε, ποτέ δεν θα σας πούν ε, ότι δεν έχουν παρουσία στη Βοσνία Το αντίθετο συναντιούνται με τον πρόεδρο Ντόντικ ε, πάντοτε κάποιες ώρες πριν από σημαντικές στιγμές και ιδιαίτερα πριν από τις εκλογές. Και μάλλον το ίδιο θα κάνουν και φέτος ο Ερντογάν. Βρήκε επιτέλους ένα τόπο στην Ευρώπη για να υλοποιήσει τη δική του εκστρατεία. Έτσι λοιπόν, Τούρκοι και Ρώσοι αναγνωρίζουν ανοιχτά ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ από τη χώρα αυτή, για τη χώρα αυτή και θέλουν να επηρεάσουν είναι μοίρα είπε πεπρωμένων τη Βοσνία Ερτσεκοβίνη. Ενώ οι χώρε του κόλπου δεν λένε ποτέ ότι είναι εκεί, αν και έχουν παρουσία. Πριν κάποιου μήνε πήγα στη Σαουδική Αραβία και έθεσα άμεσα την ερώτηση, γιατί όλοι συζητούν για αυτό το θέμα και μου είπαν οι αδερφέ, Όχι, ποτέ εμεί δεν είμαστε εκεί, δεν έχουμε παρουσία εκεί. Η Βοσνία είναι μια χώρα όπω οι άλλε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των κρατών και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν προσπαθούμε να αντιδράσουμε. Είναι ένα σημαντικό σημείο λοιπόν. Είμαι πεισμένο ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θα παρουσιάσουν τροπολογίες και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας να συνεργαστώ με όλες τις πολιτικές ομάδες για να βρούμε μια κατάλληλη διατύπωση για τη χώρα, μια χρήσιμη διατύπωση. Σε λίγο καιρό είναι και εκλογές, περίπου σε ένα μήνα και θα επεξεργόμαστε και τι δικέ μα τροπολογίε κατά τη διάρκεια τη προεκλογική ε, διαδικασία, αλλά ίσω και μετά τι εκλογέ. Ελπίζω αυτό το μετά να είναι πολύ σύντομο και να μα επιτρέψει να έχουμε και θετικά μηνύματα μετά τι εκλογέ, όχι μόνο πριν. Τώρα, για όσα υπόθηκαν από τον συνάδελφο Ράντο. Αλλά και από την κυρία Ζόφκο για την εκλογική νομοθεσία και την εκπροσώπηση. Εγώ πριν την τρίτη έκθεση του προηγούμενου έτους είπα ότι ως προς τα εκλογικά ζητήματα θα πρέπει η Βοσνία να ακολουθήσει αυτά που δέχονται και τα ευρωπαϊκά κράτη ως εκλογική μεταρρύθμιση. Και υπάρχει και νομοδότηση της Επιτροπής Βενετίας που λέει ότι κάθε τροποποίηση του εκλογικού νόμου θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Είναι κάτι πολύ λογικό θα έλεγα και ιδίω από τους σκοπιά των εκλογικών κομμάτων. Γιατί αν ένα έτος πριν τις εκλογές αλλάξεις ε, τον εκλογικό νόμο, έχεις χρόνο να εργαστείς ε, βάσει της νέας νομοθετικής πραγματικότητας. Ενώ αν το κάνεις κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες ακόμη πριν από τις εκλογές, αυτό μπορεί να ε, ταράξει και τη ζωή των κομμάτων αλλά και των πολιτών. Έδωσα αυτή τη μικρή συμβουλή όταν ήμουν στη Βοσνία Ζεγοβίνη, ε, από το 2016 ήδη, σε όλους ε, τους πολιτικούς πρωταγωνιστές ε, που συνάντησα, του είπα, θα είναι κάτι πολύ θετικό αν φτάσετε σε συμφωνία για τον εκλογικό νόμο, αλλά κάντε το γρήγορα. Ήταν αδύνατον. Και εδώ η Βόσνη είναι αδύνατο να κάνουμε μια συμφωνία, επομένως εμείς δεν έχουμε καμία εξουσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουν οι Βόσνοι. δεν μπορούμε να παρέμβουμε ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πούμε αυτό είναι ο νόμος. Δεν ε, είμαστε αυτοκρατορία εδώ. Είμαστε μια κοινότητα που θέλει κάποια μέρα να γίνει κράτος μέλος η Βοσνία Τζεγοβίνη. Λυπάμαι πολύ για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στον εκλογικό νόμο ως προς την εκπροσώπηση, όμως είχαμε πολύ καλές προθέσεις. Βέβαια δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Ε, τώρα για την ε, ομοσπονδιοποίηση που αναφέρθηκε από την κυρία Τσουίτσα, την ε, αναφέραμε στην προηγούμενη έκθεση, δυστυχώς δεν βοήθησε καθόλου. Εκ νέου, Είμαστε πολύ γενναιόδοροι. Αναφέραμε πολλές πολιτικές αρχές που ισχύουν σε διάφορα κράτη-μέλη και την αρχή της Ομοσπονδίας, του Ομοσπονδικού χαρακτήρα, όμως ε, δυστυχώς ε, δεν ε, επηρέασε καθόλου τις πολιτικές δυνάμεις της Βοζίνης τη αυτού τους. Κάναμε κάποιες προτάσεις και πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Προτείναμε μια σειρά άρχων Όμως αυτό δεν τους βοήθησε. Λυπούμαστε γι' αυτό, όμως τι μπορούμε να κάνουμε. Κάποιες μέρες ε, πριν από τις σημαντικές αυτές εκλογές, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Κριστιαν. Και καθώς έχουμε ακόμη χρόνο, ε, σου επέτρεψα να μακρηγορήσεις. Γιατί, Κριστίνη, θα έχουμε πάρα πολλέ ε, περιπτώσει να συζητήσουμε, πολλέ ευκαιρίε να συζητήσουμε την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή μια χώρα που είναι πάντοτε στο νου μα και παρουσιάζει ιδιαίτερε προκλήσει. Τώρα, η τροπολογία θέση τροπολογιών είναι 10 Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο να προετοιμάσουμε τι πρωτολογίε και πιστεύω ότι πολλοί από εσά το πράξετε. Η δεύτερη εξέταση τη έκθεση θα γίνει στι 5 Νοεμβρίου και κατόπιν η ψηφοφορία στι 20 ή στι 21 Νοεμβρίου. Ωραία, καλή τύχη στην επίσκεψή σου στο Σεράγεβο. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Μια κοινή συζήτηση για τα σημεία 7 και 8, σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική δράση για τη Συνολική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία Κερζυγία και Πρωτόκολλο Συμφωνία για σύνοψη εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κρατών μελών του αφενός και τη Δημοκρατία τη Κυρζηγία, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω. ελπίζω ότι είναι παρόντε όλοι οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την Κυρκυζία. Και τώρα θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον συγητή και για τους δύο φακέλους των μοναδικών των κριστίων Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, να σταθώ στα δύο σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντο ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Γυρίζια και έχουμε τα σημεία σε διάταξη. Επιτρέπουν μια ανανέωση τη συμφωνία που έχουμε με την Κυριαζία για την προσχω... μετά την προσχώρηση τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο σύσταση που προτείνω δείχνει ότι προφανώ και συμφωνούμε με αυτή την επικαιροποίηση. Το δεύτερο σημείο που αφορά τη συνεργασία μα με την Κυριαζία υπερβαίνει μόνο την απλή επικαιροποίηση και προτείνω να εξετάσουμε το μέλλον των σχέσεών μας. Η πρόθεση του σχεδίου έκθεσης που προτείνω είναι να συμβάλλουμε στις διαπραγματεύσεις για μια ε, σφαιρική και συνολική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερικηζίας. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε αρκετά νωρί ω Κοινοβούλιο την ε, οπτική μα γωνία σε αυτέ τι διαπραγματεύσει, γιατί ε, θεωρώ ότι ε, έχουμε αδιαφεσβήτα ένα ρόλο να διδερματίσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ε, δεν πρέπει απλώς να εγκρίνουμε, να απορρίψουμε τις συμφωνίες που μας προτείνουν. Πρέπει να συμβάλλουμε στη διαμορφωσή τους. Και για τη συμφωνία αυτή που την χάνει πραγμάτευση για την Κυριαζία είμαστε σαφείς. Ξεκάθαρα υποστηρίζουμε την εμβάθυνση των σχέσεών μας με αυτή τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο στο σχέδιο έκθεσης έχω σκιαγραφίσει ορισμένες, ε, ορισμένους στόχους που θεωρώ πολύ σημαντικούς. Πρώτον, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας οικονομίας αγοράς που θα, θα έχει σημαντικά και απτά ωφέλη ε, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για τους πολίτες. Μετά, θα πρέπει αυτή η συμφωνία να συμβάλλει στην ενίσχυση των κανόνων του ανταγωνισμού και μέσω διαφανών θεσμών. Επίσης, μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να συμβάλλει ε, την πολυμέρεια, την ε, διεθνή συνεργασία για ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Τέταρτον, στο επίκεντρο της Συμφωνία θα πρέπει να υπάρχει σαφής ε, δέσμευση σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές αξίες και τον σεβασμό των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ε, θέτω τρεις ξεκάθαρους και διακριτούς άξονες. Πρώτον, ε, συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυργιζίας στα διεθνή φόρα επισημαίνω τη σημασία της συμφωνίας για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας και μιλώ και για τη βελτίωση συντονισμού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυργιζίας στα διεθνή φόρα όπως ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ο δεύτερος άξονας, θεσμικές ε, πλευρές. Εδώ μιλώ για την ε, συμφωνία της ενίσχυσης της συμφωνίας, όπως είναι η δικαστική συνεργασία, ε, δικαιώματα του ανθρώπου. Επισημαίνω τη σημασία ενίσχυσης ε, του ρόλου ε, της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Νέας Συμφωνίας για να υπάρξει σημαντική και αποτελεσματική παρακολούθηση των συστάσεων που γίνονται παραπάνω. Και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με τα σημεία κοινού ενδιαφέροντος και κοινών συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυργιζίας. Αφενός, συνεργασία σε ζητήματα δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική λοιπόν δραστηριότητα θα πρέπει να ε, υπάρχει πολυμέρεια και δημοκρατικές αξίες. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει και ε, οικονομικά και τεχνικά και με όποιον τρόπο μπορεί αυτή την προσπάθεια. υπήρξαν και συνταγματικές ε, τροποποιήσεις το 2016. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Αυτές τι πραγματεύσει λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε το ζήτημα ε, της αξιοποίησης της δικαιοσύνης ε, και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης. Πρέπει να βασιζόμαστε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Άλλο τέτοιο σημείο έχει να κάνει με την περιφερειακή εφαρμογή της συμφωνίας στην Κεντρική Ασία. Είναι σημαντικό να επωφεληθούμε αυτών των διαπραγματεύσεων για να ενθαρρύνουμε την ε, συμβουλευτική συνεργασία και να ε, απαλύνουμε κάπως ε, τον οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ της Κυργιζίας και του Καζακστάν και του Ουσμπεκιστάν. Δύο χώρες που θα επισκεφθούμε ως Επιτροπή Εξωτερικών υποθέσεων μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτοί είναι λοιπόν οι τρεις άξονες ε, που διέπουν το σχέδιο έκθεσης. Ε, θα υποβάλω και δικές μου τροπολογίες που θα συμπληρώσουν και θα επεξηγήσουν ε, την πρότασή μου και ελπίζω να ληφθούν υπόψη αυτή την συζήτηση και κλείνοντας χαιρετίζω και καλωσορίζω τον πρέσβη της Κυριαζίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μαζί μας. Τον ε, καλωσορίζουμε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κριστιαν. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για την Κεντρική Ασία, κυρία Πέτερσεν. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Κυριαζία είναι μια μικρή νησίδα δημοκρατίας ε, στην Κεντρική Ασία. Βεβαίως ε, είναι μια αδύναμη δημοκρατία και χρειάζεται τη στήριξή μας σε κυριαρχία ε, σε πολλά επίπεδα. Οικονομικό, εμπορικό, στον τομέα της εκπαίδευσης, στην ενδυνάμωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, του κρατούς δικαίου. Αυτή η συμφωνία θα είναι μια πολύ καλή αφετηρία για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεργιζίας και προτείνω στην Επιτροπή να αποδεχτεί αυτές τις νέες τροποποιήσεις στη συμφωνία και επιβλέπω σε στενότερη συνεργασία στο μέλλον μεταξύ όλων των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Κατάλογος ομιλητών τώρα. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Ωραία, κυρία Αλιού Μαγή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ αρχικά τον ε, Κριστιαν που όπως πάντα ε, εκπονεί εκθέσεις που είναι ιδιαίτερα ακριβεί και ενδιαφέρουσες. Πριν από μερικά χρόνια πήγα στην Κυριαζία και πρέπει να πω ότι αυτό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι βλέπω ότι ακολουθούμε ε, το ίδιο pattern ε, στις συμφωνίες, ανεξάρτητα από το ποια είναι η χώρα. Και αυτό μου φαίνεται λίγο παράδοξο, γιατί βλέπουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο συμφωνίες, με τις ίδιες διατυπώσεις, με τις ίδιες παραπομπές. Σε χώρες όπως ε, το Μαρόκο μέχρι σε χώρες όπως η Κυργυζία. Είναι σημαντικό εδώ να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες μνήες και επισημάνσεις ε, που θα αντικατοπτρίζουν τις χώρες αυτές, ε, την αφετηρία τους και το που βρίσκονται σήμερα. Και αυτό πρέπει να γίνεται με πολύ συγκεκριμένο, προσδιορισμένο και ρεαλιστικό τρόπο. Δεύτερον, αυτός ο τύπος συμφωνίας δεν μπορεί να διακρίνεται, όπως είπε και ο Κριστιαν, από ένα σύνολο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τελικά ένα όραμα των σχέσεων που θέλει να διαμορφώσει με αυτές τις χώρες. Τη στιγμή που η Κίνα ε, δημιουργεί μια νέα διεθνή πολιτική για τον νέο δρόμο του μεταξιού, εμείς ως Ευρωπαίοι τι όραμα έχουμε να αντιπροβάλλουμε για το σύνολο αυτών των χωρών που έχουν και σημαντικό πολιτισμό, αλλά και είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον ε, της οικονομίας και του εμπορίου μας. Αφενός λοιπόν θα πρέπει να εξετάζουμε και αυτή τη στιγμή αγνοούμε και την πραγματικότητα της κάθε χώρας, αλλά αγνοούμε και παραμελούμε και την ευρύτερη εικόνα. Τι κάνουμε τελικά με την Κεντρική Ασία, πέραν της υπογραφής ε, επιμέρους ε, συμφωνιών. Αν θέλουμε μία νέα διεθνή πολιτική, πρέπει να αναλογιστούμε το μέλλον όλων αυτών των ε, περιφερειών. Φυσικά και διαφέρει μία χώρα από την άλλη, αλλά είναι μία περιφέρεια που δεν ε, ε, γίνεται να την παραγωνίσουμε, να την αμελήσουμε. Ξέρω ότι μια τέτοια συμφωνία δεν ε, μας επιτρέπει να τα αναφέρουμε όλα αυτά σε μεγαλύτερο βάθος, αλλά στις παρουσιάσεις του θα ήθελα να παρακαλέσω τον Κριστιαν να αναφέρει ότι η Ευρώπη θα πρέπει, μπορεί και πρέπει να έχει μια οικονομική ε, και στρατηγική φιλοδοξία για αυτές τις περιφέρειες. Ευχαριστούμε πολύ, Μισελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα η σύγκριση της Κυριαζίας με το Τατζικιστάν ή το Ουσβεκιστάν ή ακόμη και το Τουρκμενιστάν ε, είναι ε, κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση στην Κυριαζία από όλες αυτές τις χώρες, όμως ε, σίγουρα δεν είναι καιρόδυνα τα πράγματα και έχουμε μία τάση να πιστεύουμε ότι καθώς ε, υπάρχει μία υπερδομή ότι αυτή σηματεύει και τη δομή. Όμως δεν είναι βέβαιο αν δεν καταλαβούμε ποια είναι ακριβώς η εύθραστη κατάσταση της κερζυγίας, όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή Είχαμε και τις σειράξεις στην κοιλάδα της Φεργάνα στο παρελθόν, που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη περιοχή και που φυσικά πλήττουν το Τζατζικιστάν και το Κυργιστάν και να μην μιλήσουμε και για την επιρροή του Αφγανιστάν με ε, όλες αυτές ε, τις... Ε, την εμπορία, το εμπορίο ναρκωτικών ε, στην ε, περιοχή, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για να τα κατανοήσουμε. Επίση πρέπει να κατανοήσουμε σε ποια θέση βρίσκεται η Κυργυζία. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της βόρεια ε, και περιοχής, του Μπισκέκ και του Νότου, που είναι μια πιο αγροτική περιοχή, αλλά στην πόλη του Όσου, το χάρη, έχουμε περισσότερους Ουσμπέκου παρά Κυργίζιου. Αυτό είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη υπόψη για να καταλάβουμε και τις διάφορες ε, υπεδρομές ε, των κομμάτων ε, Αναλόγω αν η βιβάση του εκλογή είναι περισσότερο στο βορρά ή το νότο και πρέπει να δούμε και ποια είναι η θεμελιώδη διαφορά που υπάρχει μεταξύ κράτου και κοινωνία στην Και Γιατί, Γιατί η κοινωνία ε, πιστεύεται πολύ περισσότερο στου αξαλάξ, στι λευκέ γενιάδε, στου περίφημου σοφού που δημιουργούν τα συμβούλια. Και σε αυτά τα συμβούλια επιλύονται ζητήματα ε, που είναι σημαντικά και ποινικά αλλά και αστικά θέματα. Αυτό γιατί, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς και γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί οι κρατικοί θεσμοί έχουν ε, πολύ μεγάλη παρουσία. Ε, κάποιο φορά που είναι ε, παίρνει τη διαφθοράς που είναι ο κοινός παρανομαστής στην περιοχή και η δικαιοσύνη ε, ουσιαστικά εξαρτάται πάρα πολύ από τις πραγματικές εξουσίες ε, και από τις πολιτικές αλλά και τις οικονομικές εξουσίες. Πρέπει το χάρη. Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπλικανικό Κόμμα, έχει ως ηγέτη τον κύριο Παπάλοφ που είναι ένας ολιγάρχης. Αυτά είναι σημαντικά. Όταν το εμπόριο μπαίνει στην πολιτική, ε, σημαίνει ότι η πολιτική αποτελεί συνέχεια ε, του εμπορίου. Αυτά όλα είναι σημαντικότατα και θα πρέπει ε, πέρα από την ιστορική συμφωνία θα πρέπει να κατανοήσουμε τι υπάρχει και κάτω από το κέλυφος, ποια είναι η ουσία της χώρας και σε τι συνίσταται ο πληθυσμός. Ευχαριστώ. Περνάμε στην κυρία Αντικίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω τις διαπραγματεύσει για μια νέα εξχρονισμένη συμφωνία που θα επικαιροποιήσει το PCA του 1999. Ε, Είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε μια πετυχημένη και ισορροπημένη συμφωνία δεύτερης γενιάς. Ταυτόχρονα όμως θέλω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι θα πρέπει να, να εντοπίσουμε ποια είναι η θέση της στην ε, κεντρική ε, Ασία. Θα πρέπει να είναι η βάση αυτή για δομημένους στόχους και στρατηγικές για το Κυρκιστάν. Συγκεκριμένα είναι σημαντικό σε παγκόσμιο πλαίσιο να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και την Κίνα ε, χώρες τις οποίες το Κυρκιστάν βλέπει στρατηγικούς εταίρους. Στις 6 Ιουνίου η Κίνα και το Κυργιστάν αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Αν αφήσουμε την περιοχή αποκλειστικά στη Ρωσία και στην Κίνα, αυτό θα έχει πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Θα πρέπει να, υπάρξουν, ναι, υπάρξει μια νέα συμφωνία με όρους που θα φορούν ε, την οικονομία, το εμπόριο, την ε, χρηστή διακυβέρνηση και το δίκαιο, το κράτος δικαίου αν θέλουμε να έχουμε έναν εταίρο ε, στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, κανολόγιο του Κυργιστάν, τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει διατάξει και δεσμεύσει στη νέα συμφωνία για την δημοκρατία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δημιουργία όρων για ε, δίκαιο εμπόριο. Όλα αυτά πρέπει να είναι αναπόσπαστα ε, κομμάτια της νέας συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Λοιπόν. Ο λόγος στην κυρία Πέτρα Γκασπάρβα από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που είναι υπεύθυνη για το Κυργιστάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνεται να συμμετάσχω στον διάλογο. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία από την πλευρά μου για τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τη 19η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Οι σχέσεις μας έχουν ε, εξελιχθεί δυναμικά τα τελευταία δύο χρόνια με το Κυργιστάν και υπάρχει ανάγκη μια νέα συμφωνία εξχρονισμένη να αντικαταστήσει την παλιά συμφωνία της δεκαετίας του 90 όχι μόνο επειδή το Κυργιστάν έχει εξελιχθεί σημαντικά είναι η χώρα που έχει προδεύσει περισσότερο όσον αφορά ε, τη διακυβέρνηση, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης έχουμε πρόοδο στις οικονομικές σχέσεις. Με την συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο συνεργαζόμαστε εντατικά στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις καθώς και τις μεταρρυθμίσεις ε, στο δικαστικό σύστημα, στην εκπαίδευση και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η νέα συμφωνία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε τους τομείς στους οποίους συνεργαζόμαστε. Θα υπάρξουν νέοι τομείς συνεργασίας όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία δεν ήταν πολύ ψηλά στο θεματολόγιο στην δεκαετία του 90, αλλά θα περιλαμβάνει και τομεί στου οποίου έχουμε ήδη συνεργαστεί, χωρίς όμως να έχουμε τη νομική βάση, όπως είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η Συμφωνία Νέας Γενιάς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει όλα αυτά που αναφέρονται εδώ από τους ε, αντιπροσώπους για, την, ε, για τις αλλαγές στην περιοχή, Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή ε, στις νέε στρατηγικέ ε, για την Κεντρική Ασία. Λαμβάνουμε υπόψη τι παγκόσμιε εξελίξεις, αλλά την παγκόσμια στρατηγική και τις νέες στρατηγικές για το Αφγανιστάν και την στρατηγική συνδεσιμότητας. Άρα δεν βλέπουμε τον Κυριστάνο ως ένα ξεχωριστό κομμάτι, μια ξεχωριστή χώρα. Βλέπουμε την περιφέρεια σαν σύνολο για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη σύγκληση των διεθνών προτύπων και συγκεκριμένα αναφορικά με την Ρωσία και την Κίνα της οποίας αναφέρατε. Μέχρι στιγμής έχουμε την νέα στρατηγική και την νέα συμφωνία που θα πρέπει να αποτελέσουν όχι μόνο για να εφαρμόσουμε το όραμά μας το πολιτικό και το στρατηγικό στην περιοχή. Μέχρι στιγμής είχαμε τέσσερις γύρους πραγματεύσεων από τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Ο επόμενος γύρος είναι τον Οκτώβριο. Βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον και προσπάθεια και πολιτική βούληση από την πλευρά των εταίρων μας στο Κυριστάν. Και εμείς από την πλευρά μας είμαστε δεσμευμένοι να προχωρήσουμε γρήγορα και να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη ε, συμφωνία για τα επόμενα 20 χρόνια. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο Κρίστιαν Πρέντα θέλει να συνοψίσει. Όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους. Χρονοδιάγραμμα. Υποβολή τροπολογιών σε δύο μέρες. 31η, με συγχωρείτε, έχουμε νέα προθεσμία 5η Σεπτεμβρίου, αντί 29η Αυγούστου. Η με συγχωρειτε εχουμε νεα προθεσμια 5 η σεπτεμβριου 29 η αυγουστου η ψηφοφορια στην ΑΦΕΔ 8 ή 9 Οκτωβρίου ή στην 22 Νοεμβρίου και θα φτάσουμε στην Ολομέλεια μέχρι τα Χριστούγεννα, ευελπιστούμε. Αυτά για Προς το παρόν θα συνεχίσουμε τις συνεδρίσεις στις 2.30. Ε, θα γίνεται αλλαγή απόψεων με τον νέο επικεφαλής ε, της ε, αποστολής της Αφρίξης στην Λιβύη. Ευχαριστώ.